Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων. Ανοιχτή σε όλους τους βουλευτές και χαίρομαι που βλέπω τόσους συναδέλφους εδώ παρόντες. Ε, κυρίες και κύριοι, θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Βαρόμπαϊ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον κύριο Μπαρόσο, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα όσο και σημαντική η σημερινή συνεδρίαση. Θα μας ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των ε, συνεδριάσεων ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22 του μηνός. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Βάρον Πέι, Πρόεδρο του Συμβουλίου. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να μας ενημερώσετε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτές, ε, την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν σύντομο αλλά αποτελεσματικό και αποδοτικό. Ήταν μια ευκαιρία για τους Ευρωπαίους ηγέτες να αφιερώσουν χρόνο στη τομέα της ενέργειας. Επίσης δόθηκε νέα όθηση σε θέματα που για πολύ καιρό είχαν παγώσει, ιδιαίτερα όσον αφορά την φοροδιαφυγή και τις ε, φοροαπάτες. Ε, επίσης, ε, είχαμε και μια συνεδρίαση για την κρίση, την οποία πια έχουμε συνηθίσει. Βέβαια, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα, αλλά είμαστε στη σωστή πορεία. Να αρχίσουμε με την ενέργεια, πώς αυτό επηρεάζει τους καταναλωτές μας και τις οικονομίες μας. Από την τελευταία διάσκεψη κορυφής που είχε αφιερωθεί στην ενέργεια, το Φεβρουάριο του 2011, έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, έκαναν βήματα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας και από κοινού με το Συμβούλιο υιοθετήσαμε την οδηγία περί επάρκειας σε ενέργεια που θα μας επιτύχει να επιτύχουμε ε, τον στόχο του επάρκειας ενέργεια του 20% μέχρι το 2020. Ταυτόχρονα από το 2011 έχει αλλάξει ο κόσμος. Όπως ένας από τους ηγέτες είπε, είμαστε τώρα στα μέσα μιας παγκόσμιας ενεργειακής επανάστασης θα φτάνει κανείς να δει πέρα από τον Ατλαντικό για να δει ότι αυτό αληθεύει. Έχουμε αναζητήσει νέους πόρους, αυξάνονται όμως οι τιμές και σύντομα η Ευρώπη θα είναι η μόνη ήπειρος που θα εξαρτάται ε, από την εισαγόμενη ενέργεια. Ειλικρινά δεν είναι πολύ άνετη αυτή η κατάσταση για μας, όχι για τα νοικοκυριά μας που αισθάνονται το βάρος των ψηλών τιμών ενέργειας και γι' αυτό και ε, το ενδιαφέρον μας στα δικαιώματα του καταναλωτή ήταν κεντρικό, αλλά το ίδιο δύσκολο είναι και για την την ε, βιομηχανία μας που πολύ συχνά πληρώνει διπλά για τον ηλεκτρισμό. Όμως θέλουμε να κρατήσουμε τα εργοστάσια και τις θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη. Οπότε η προσιτή και η βιώσιμη ενέργεια είναι πολύ βασική. Εμείς στην Ευρώπη δεν, όμως, δεν προβλέπουμε κάποια βασική αλλαγή στον ορίζοντα. Υπήρχε επίσης συνένεση, ε, ε, που αντικατοπτρίζεται και στα πορίσματα του Συμβουλίου ότι χρειάζεται μια κοινή προσέγγιση και όχι 28 χωριστέ προσεγγίσεις. Μια κοινή προσέγγιση που θα, αποτελείται, θα βασίζεται σε τέσσερα σημεία. Καταρχήν, επάρκεια ενέργεια. Η υιοθέτηση, όπω είπα, της οδηγίας περί επάρκεια ενέργεια έδωσε πραγματική όθηση. Τώρα η πρόκληση είναι η εφαρμογή τη γιατί ε, η φθηνότερη και η καθαρότερη ε, ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Να δημιουργηθεί μια πραγματική ε, ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Οι ηγέτες επέμειναν για την πρόοδο πέρα από την μάλλον νωρίτερα από την προθεσμία του 2014 και την προθεσμία του 2015 για τις διασυνδέσεις. Τονίστηκε η ανάγκη να διασυνδεθούν καλύτερα οι υποδομές ενέργειας και αυτό αντικατοπτρίζεται επίση στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Όμως γι' αυτό, και αυτή είναι η τρίτη μου προτεραιότητα, χρειάζονται επενδύσεις. Όχι κάτω από ένα τρισεκατομμύριο μέχρι το 2020 σε σύγχρονες υποδομές αλλά και στην έρευνα και την ανάπτυξη. Η διευκόλυνση για τη σύνδεση της Ευρώπης παίζει σημαντικό ρόλο εδώ για να φτάσουμε σε ταχεία συμφωνία για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμως ένα μεγάλο μέρος των μελλοντικών επενδύσεων θα πρέπει να προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο, το να Για να μπορέσουν να δαπανίσουν οι επενδυτέ, θα πρέπει να γνωρίζουν περίπου πού σκοπεύουμε να βρισκόμαστε σε 20 με 30 χρόνια. Πιο προβλέψιμη πολιτική δηλαδή για την ενέργεια και για το κλίμα. Ο σχεδιασμός είναι πολύ σημαντικός, αλλά είναι και πολύ ευαίσθητη η κατάσταση, όπως βλέπουμε από την ψήφο ε, για την τροπολογία για το, για το backloading με βάση το πράσινο βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο καλωσορίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ε, μέχρι το τέλος του χρόνου η Κομισιόν θα υποβάλει πιο συγκεκριμένες προτάσεις και μετά από αυτό θα δουλέψουμε για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο μέχρι το Μάρτιο του 2014 και είναι πολύ σημαντικό να, να συνεχίσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες εντωμεταξύ. Τέταρτη προτεραιότητα, η διαφοροποίηση των πηγών ενέργεια. Τα κράτη-μέλη που καταφέρνουν να μειώσουν την εξάρτησή του από έναν μόνο προμηθευτή ή μόνο μία συγκεκριμένη διαδρομή προμήθεια βλέπουν τα ωφέλη τη διαφοροποίηση. Και η πρόκληση είναι σαφή. Η Ευρώπη πρέπει να εκμεταλλευτεί το ενεργειακό τη δυναμικό πλήρω ε, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, που είναι και μεγάλη πηγή θέσεων απασχόληση, αλλά και αναπτύσσοντα ασφαλεί και βιώσιμου τρόπου για να ε, εκμεταλλευτεί εκμεταλλευτεί συμβατικούς και μη ε, πόρους ή πηγές. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και κατάλληλη χρήση του αερίου σχιστόλιθου. Ε, η Κομισιόν θα αξιολογήσει την κατάσταση αυτή και φυσικά αναγνωρίζεται ρητά στη συνθήκη ότι εξαρτάται από την κάθε χώρα να αποφασίσει για το μείγμα ενέργειας που θα χρησιμοποιήσει. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό μήνυμα το ότι από κοινού συμφωνήσαμε για αυτά τα τέσσερα σημεία. Τώρα χρειάζεται επιγόντως να δοθεί συνέχεια σε αυτά που αποφάσισαν οι ηγέτες και γι' αυτό και στα συμπεράσματα τονίζουμε την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό και προηγούμενο συντονισμό για τα, τις ε, μεγάλες εθνικές αποφάσεις περί ενέργειας με ενημέρωση και στις άλλες χώρες. Καλό η κυλιόμενη Προεδρία να το μεταφράσει αυτό σε συγκεκριμένη δράση στο, επίπεδο, στο υπουργικό επίπεδο. Και ζητάμε από την Κομισιόν να αναλύσει τις τιμές και τον αντίκτυπο στα νοικοκυριά μέχρι το τέλος του έτους, ούτως ώστε αυτά τα στοιχεία να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν άλλες ε, άλλα θεματικά ευρωπαϊκά συμβούλια που είναι προσχεδιασμένα και τα περισσότερα από αυτά εξάλλου σχετίζονται και με το θέμα του ανταγωνισμού. Και αποφασίσαμε να επανέλθουμε στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής ήδη το Δεκέμβριο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή αυτών των προσανατολισμών. Δεύτερο θέμα σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή. Δεν είναι νέο θέμα και σίγουρα είναι πολύ λεπτό και ο πρόοδος εδώ είναι δύσκολη. Ωστόσο αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν διαφορετικό και γιατί διότι υπήρχε μια συνήθιστη όθηση λόγω μια σειρά σκανδάλων που ξέσπασαν σε διάφορες χώρες. Σε φάση δημοσιονομικής λιτότητας και εξυγίασης, όπου οι κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν δύσκολες αποφάσεις που επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών τους, η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή ε, γίνεται, καθίσταται ακόμα πιο απαράδεκτη από, ε, από ποτέ. Και τα ποσά είναι εντυπωσιακά, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που φεύγουν, που λείπουν ετησίως από την Ευρώπη. Ήταν πλέον η κατάλληλη στιγμή για να αρχίσουμε να εντείνουμε τον αγώνα και γι' αυτό και ε, βάλα αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Από τη φύση της η φοροδιαφυγή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λύσει, ένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει μια χώρα μόνη της. Και παρότι είναι τόσο ευαίσθητο θέμα, και αντικατοπτρίζεται με στην, την ομοφωνία που προβλέπεται για αυτά τα θέματα στην ε, συνθήκη, δεν υπάρχει εμβολία ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την αφοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και μόνο ενωμένοι στην Ευρώπη μπορούμε να δώσουμε παγκόσμιο στο παράδειγμα. Τον Μάρτιο μόλις είχαμε θίξει το θέμα και την προοπτική μια διάσκεψη κορυφή που θα είναι αφιερωμένη στη φοροαποφυγή και στη φοροδιαφυγή. Να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση ώστε να κινηθούν τα πράγματα μετά από χρόνια τέλματος. Είμαι ευτυχής λοιπόν που το Συμβούλιο μπόρεσε να ξεμπλοκάρει πολλά παγωμένα θέματα, κίνηση, επιτάχυση με σαφείς προθεσμίες. Σήμερα είμαι ευτυχής που μπορώ να σας αναφέρω ότι υπάρχουν κάποια πρώτα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Καταρχήν η φοροαποφυγή ε, με το ΦΠΑ. Οι ηγέτες περιμένουν οι υπουργοί τους να υπογράψουν το αργότερο τον Ιονίο σε ένα σύνολο ε, μέτρων ταχείας ανταπόκρισης ε, τα κράτη να μπορούν να παρεμποδίσουν τους φοροδιαφεύγοντες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Δεύτερο σημείο, ίσως να γνωρίζετε ότι πριν δύο εβδομάδες, πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συμμετείχα για πρώτη φορά σε ένα πρωινό εργασία στο ΕΚΟΦΗΝ, όπου τόνισα στους υπουργού Οικονομικών την ανάγκη να εντατικοποιηθεί ο αγώνας μας κατά της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Πριν από δύο εβδομάδες, οι υπουργοί Οικονομικών ε, συμφώνησαν στο διαπραγματευτική εντολή αφορά τη φορολόγηση των ε, καταθέσεων, Αποφάσισαν να αρχίσουν αμέσω διαπραγματεύσεις με την, Ελβετία, το Λιχτεστάιν, ε, το Σαν Μαρίνο ώστε αυτές οι χώρες να χρησιμοποιήσουν πλέον κοινέ προδιαγραφές επί τη βάση της αναθεωρημένης οδηγίας περί ε, ε, φορολόγησης των αποταμιεύσεων. Αυτό σημαίνει ενωσιακή συνένεση όσον αφορά μια ενιαία φορολόγηση και αυτό είναι ένα συμπέρασμα όπου περιλαμβάνεται και η προθεσμία περί του τέλους του έτους. Τρίτο σημείο που συνδέεται, θέλουμε όλη η Ένωση να πιέσει για να τεθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές παγκοσμίω για την ανταλλαγή πληροφοριών για τα θέματα φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και εμείς προωθούμε την υιοθέτηση τέτοιων παγκοσμίων προδιαγραφών. Μια ομάδα κρατών μελών ξεκίνησε αυτή τη δράση και τώρα πλέον είναι αποδεκτή σε νοσιακό επίπεδο. Θα πρέπει να τονίσω δε ότι αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών υπάρχει ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά χρειάζεται να ενισχυθεί και να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογή της. Η, οδηγία, η αναθεωρημένη οδηγία για τις ε, αποταμιεύσεις και η αναθεωρημένη οδηγία για την ε, φορολόγησή τους θα προβλέψουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ε, εφοριών των κρατών μελών. Τέταρτο σημείο, πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων φορολογικό σχεδιασμό επιθετικό ή φοροδιαφύγη από τι εταιρείε κτλ. χρειάζεται ενία ε, πανευρωπαϊκή προσέγγιση. Συμφωνήσαμε και θέσαμε προθεσμίε μέχρι τα τέλη του έτου, για παράδειγμα, για αναθεώρηση ε, των θεμάτων που αφορούν την ε, επικουρικότητα και τις οδηγίες για ε, την ομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θα επανέλθουμε ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τέλος, σύντομα, συζητήσαμε και την κατάσταση στη Συρία. Διατρανώσαμε και πάλι την προσήλωσή μας σε μια πολιτική λύση. Δώσαμε την υποστήριξή μας σε μια πρωτοβουλία διεθνούς διασκέψεως βάσει των ε, αρχών που θεσπίστηκαν στην Γενέβη τον Ιούνιο του 2012. Ε, ζητήσαμε από τους Υπουργούς Εξωτερικών να προετοιμάσουν ε, τη διάσκεψη και να σχεδιάσουν ένα νέο σύστημα κυρώσεων για το παλιό εκπνέει 1η Ιουνίου του 2013. Καλή Ευρωπαϊκή Ένωση για πολιτική λύση της σύραξης και καλωσορίζουμε την διεθνή διάσκεψη. Το Συμβούλιο επέκτηνε, παρέτεινε κατά 12 μήνες όλα τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα με εξαίρεση του αποκλεισμού του εμπάργου στα όπλα. Είναι πολύ σημαντικό να καθοδηγήσουμε τις εθνικές πολιτικές. Επίσης συμφώνησε το Συμβούλιο ότι τα κράτη-μέλη επί του παρόντος δεν θα προχωρήσουν ε, στην παροχή ε, όπλων. Ε, αποφάσισαν οι Υπουργοί ότι πριν την 1η Αυγούστου θα επανέλθουν σε αυτό το θέμα μετά από έκθεση που θα καταθέσει η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος ε, σχετικά με την έκβαση των συνομιλιών της Γενέβης. Σε τελική ανάλυση λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πολλά θέματα αποφασίστηκαν με πολλές προθεσμίες και δρομολογήθηκαν στο Συμβούλιο. Και συμπίπτει να γίνεται αυτό ακριβώς ένα χρόνο πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών εκλογών. Ένας ακόμα λόγος για να είμαστε όλοι προσιλωμένοι σε αυτές τις υποθέσεις. Ε, πριν τελειώσω θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας άλλη μια σκέψη για ένα θέμα που έθεσε ο πρόεδρός σας, ο κύριος Σούλτς, που είναι η ενεργεία των νέων. Στην επόμενη συνεδρίασή μας, τον Ιούνιο, ε, θα θέσουμε την καταπολέμηση της ενέργειας των νέων υψηλά στις προτεραιότητες. Αυτό το συμβούλιο θα είναι μια ε, προσπάθεια και μια ευκαιρία να κινητοποιηθούμε όλοι προς ένα κοινό στόχο, να δώσουμε στους νέους τις εγγυήσεις ότι θα έχουν είτε εκπαίδευση, άσκηση, μετακπαίδευση ή ε, απασχόληση εντός τεσσάρων μηνών από την αποφύτισή τους. Αυτό εγκρίθηκε στις 22 Απριλίου σε σύσταση του Συμβουλίου. Τις τελευταίες ημέρες διάφορα κράτη-μέλη ανακοίνωσαν ότι θα προχωρήσουν ε, με υποβολή ιδεών για ε, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών υπέρ τη απασχόληση των νέων. Καλωσορίζω και ενθαρρύνω αυτέ τι πρωτοβουλίε. Την Παρασκευή απέστειλα επιστολή στα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου τα καλώ να μοιραστούμε ιδέε και να δραστηριοποιηθούν εν ώψη του Συμβουλίου του Ιουνίου. Επίση, στην επιστολή μου. απευθύνθηκα και στους κοινωνικούς εταίρους να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έχει θέσει ως προτεραιότητα την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων με 6 δισεκατομμύρια που ε, αφιερώνονται στην αντίστοιχη πρωτοβουλία για τους νέους ε, στην πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι μέχρι πρώτου του 2014 θα είναι έτοιμο και πλήρως επιχειρησιακό αυτό το πρόγραμμα. Χρειάζεται υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ε, πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των προσδοκιών πολλών νέων που περιμένουν πολιτική δράση από μας. Ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε πολλές υποχρεώσεις αναλάβει μέχρι τα τέλη του έτους. Να δούμε τι θα μας πει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα, ο κύριος Δουράου Παρόσο, να μας δώσει τη δική του ε, θεώρηση και εκδοχή των ε, πεπραγμένων της περασμένης εβδομάδας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε και κύριοι. Ήταν πολύ επαγγελματικό το συμβούλιο αυτό και δεν είχε τόσο δραματικές εξελίξεις αντίθετα από άλλα. Ωστόσο, τα θέματα έρονται στο ύψος των προκλήσεων και πάμε στη σωστή κατεύθυνση και σε ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική, δηλαδή κάνουμε βήματα προς την κατεύθυνση μιας πιο ολοκληρωμένης, αποτελεσματικής, αποδοτικής και φιλικής στον καταναλωτή ευρωπαϊκής ε, αγοράς ενέργειας και το σωστό μείγμα. Επίσης, ε, καλά τα πάμε και για θέματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και των φορολογικών απατών. Αλλάζουμε δηλαδή το πλαίσιο έτσι ώστε να συνεργάζονται οι χώρες για να κλείσουν τα διάφορα παραθυράκια και να βελτιωθούν τα πρότυπα, ώστε ο καθένας να συμβάλλει δικαίως κατά τη δύναμή του. Εγώ θα ήθελα βέβαια τα συμπεράσματα του Συμβουλίου να είναι και πιο φιλόδοξα και πιο συγκεκριμένα σε ορισμένα σημεία. Ωστόσο υπάρχει μια όθηση και κινούμαστε και στις δύο αυτές τροχές προς τα εμπρός. Τώρα βέβαια πρέπει να ακολουθήσουν οι πράξεις, η δράση, στην βάση των ε, προτάσεων που έχουν κατατεθεί και στη βάση των όσων έχουν ήδη αποφασιστεί. Κυρίε και κύριοι, ε, η συζήτηση για την ενέργεια, εγώ κατέθεσα ένα χάρτη για να στηρίξω τη συζήτηση αυτή της κατάστασης ενέργειας που αλλάζει παγκόσμια. Οι διαφορές στις τιμές και στις συνθήκες της αγοράς στις διάφορες χώρες της Ευρώπης είναι αποκαλυπτικές και σημαίνουν ότι χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία. Είναι κρίσιμη η μεγαλύτερη συνεργασία και για την ανταγωνιστικότητά μας και για την ανάπτυξή μας. Και αν πραγματικά είχαμε και ανάγκη να μας το θυμίσει κανείς πόσο απαραίτητο είναι να ολοκληρωθεί η ενεργειακή αγορά, να, τον έχουμε τώρα. Αν χρειαζόμασταν, ας πούμε, κίνητρο για να δουλέψουμε πάνω στην ενέργεια, η σύγκριση με τις εξελίξεις εκτός Ευρώπης θα πρέπει να μας αρκεί ως τέτοιο κίνητρο. Παράδειγμα, το 2012 το βιομηχανικό αέριο κόστιζε τέσσερις φορές λιγότερο στις ΗΠΑ από ό,τι στην Ευρώπη για το ηλεκτρικό ρεύμα. Η Ευρώπη είναι διπλάσια ακριβή από τις ΗΠΑ. Επίσης γίνεται αγώνας τώρα για το ποιος θα προλάβει να εξασφαλίσει τους περισσότερους πόρους. Και εκεί χάνει η Ευρώπη. Η παγκόσμια δε κατάσταση ενέργειας δεν είναι υπέρ της Ευρώπης, αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε ητοπαθείς. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Εγώ χαίρομαι λοιπόν που γενικά υποστηρίχθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα σενάριο που το λέω εγώ να μην το βάλουμε κάτω. Να αρχίσουμε τώρα να εφαρμόζουμε αποφάσεις για την πολιτική της ενέργειας που θα έχουν επιπτώσει για το μέλλον. Άρα, εδώ χρειαζόμαστε πρόοδο σε πέντε τομείς. Πρώτος, ολοκλήρωση της ενιαίας εσωτερικής δηλαδή αγοράς της ενέργειας, κατάργηση των κολλημάτων και άλλων φραγμών και ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για εταιρείε και καταναλωτές. Δεύτερο, επενδύσεις στην καινοτομία. Τρία, μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Τέσσερα, ανανεώσιμες ενέργειες να γίνουν πιο φθηνές και πιο αποδοτικές. Πέντε, διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας αναζητώντας νέες διεθνείς πηγές. Άρα προχωρούμε σε αυτά που λέμε μια βάση ας πούμε για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή κοινότητα. Εάν οι διάφορες χώρες μέλη έχουν διαφορετικά μείγματα ενέργειας, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα αν δράσουμε μαζί. Αυτό θα ευελτιώσει και την ανταγωνιστικότητά μας και την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας και βέβαια τη βιωσιμότητα. Και βέβαια τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις δεν χρειάζεται εγώ να σας υπενθυμίσω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για ε, την διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Μέσα στο πλαίσιο δηλαδή του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου, όπου υπάρχει περιθώριο για την ενέργεια. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα των προγραμμάτων αυτών. Και η πραγματική δοκιμασία δεν θα είναι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά στην εφαρμογή τους. Όλα έχουν τεθεί επιτάπητος. Πρέπει να εφαρμόσουμε τα όσα έχουν συμφωνηθεί και να δράσουμε επομένως τολμηρά. Κυρίε και κύριοι, η αντιμετώπιση των φορολογικών απατών και της φοροδιαφυγής ήταν το άλλο μεγάλο θέμα. Χαίρομαι για την ισχυρή στήριξη που προσφέρει στην προσέγγιση της Κομισιόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και στο θέμα αυτό γνωρίζουμε την έκταση του προβλήματος, γνωρίζουμε τις επιζήμες επιπτώσεις του και γνωρίζουμε και τι πρέπει να πράξουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Οι περισσότερες αναγκαίες προτάσεις έχουν κατατεθεί εδώ και καιρό. Πρόταση της Κομισιόν του 2008 για να κλείσουν τα παραθυράκια στην ε, οδηγία περί καταθέσεων. Επίσης για τη διαπραγμάτευση εντολών με για τις μάλλον διαπραγμάτευσης με ε, γειτονικέ χώρε. Αυτά έχουν ήδη προταθεί από τον προηγούμενο Δεκέμβρη. Και για τους φορολογικούς παραδείσου, πάλι από πέρσι. Και εδώ όμω οι δραματικές ζημιές που έχουμε αντιμετωπίσει δεν φαίνεται να έπεισαν αρκετά τις χώρες μέλη έτσι ώστε να οδηγηθούν σε αποφασιστικά συμπεράσματα. Τώρα επιτέλους υπάρχει, σημειώνεται μια νέα όθηση ενισχυμένη από μερικά ατυχή πούμε παραδείγματα τα οποία έφεραν στο φως της δημοσιότητας στα διάφορα μέσα. Και στη βάση αυτών εγώ ζήτησα από τους ηγέτες να προχωρήσουν. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου αναφέρονται και στην προτεραιότητα που οφείλει να δίνεται στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Αυτή δε να επεκταθεί σε όλες τις μορφές εισοδήματος και να προωθηθεί ως τα νέα διεθνή πρότυπα. Αυτό είναι σωστό. Αυτό βεβαίω είναι θετικό Παρ' όλα αυτά όμω εκφράζει τη λύπη τη η Κομισιόν διότι τελικά δεν επιτεύθηκε συμφωνία πάνω σε ξεκάθαρε πρόθεσμίε για την πλήρη εισαγωγή και εφαρμογή τη αυτομάτη ανταλλαγή πληροφοριών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί βέβαια δεν θα ανακόψουμε την ταχύτητά μα, θα υποβάλουμε την τελευταία μα πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών τι επόμενε εβδομάδε. και πριν από το επόμενο ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του τέλου Ιουνίου. Έχουμε τώρα επιτέλου την εντολή για να διαπραγματευτούμε με την Ελβετία, το Λίχτενστάιν, το Μονακό και το Σαν Μαρίνο και την αντονά. Και θα το πράξουμε αυτό εντατικά και γρήγορα. Και χαίρομαι για τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την έγκριση τη ε, οδηγία ε, καταθέσεων πριν από τέλο του χρόνου. Όλα αυτά τα βήματα είναι θετικά για του Ευρωπαίου. Πέρα από αυτά γνωρίζουμε ωστόσο ότι οι φορολογικέ απάτε και η φοροδιαφυγή είναι και παγκόσμια θέματα. Έτσι θα διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας ως Κομισιόν τις επόμενες εβδομάδες για να βελτιώσουμε την διεθνή συνεργασία και ιδίω στο G8, όπου μαζί με τον πρόεδρο του Συμβουλίου θα προσωπήσω την Ένωση τον επόμενο μήνα στη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά και στο G20 και στον ΟΟΣΑ υπήρξε πρωτοπόρο η Ευρωπαϊκή Ένωση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών και πρέπει να παραμείνει στο προσκήνιο των προσπαθειών να καθιερωθεί αυτό ω το νέο διεθνέ πρότυπο. Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα βεβαίω, τα οποία δεν θα σα αναπτύξω απαραίτητα αυτή τη στιγμή σήμερα. Είναι σημαντικά όμω σε αυτή την προσέγγιση για την καταπολέμηση τη φοροδιαφυγής και βεβαίω και, και του φορολογικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων για να αποφύγουν τη φορολόγηση. Χρειάζεται ωστόσο να γίνει Δεχτώ και, το, και δεχτεί και η αρχή της φορολογικής διαφάνειας από τις επιχειρήσεις. Σε αυτό δίνουμε εμείς προτεραιότητα. Μία κέρια ανησυχία μου που θέλω να μοιραστώ μαζί σας όταν συζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά είναι η εξή. Αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά αποτελεσματικοί και εσωτερικά αλλά και διεθνώ, δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να προχωρήσουμε όλοι μαζί και να βασιστούμε στο κοινό μα ευρωπαϊκό πλαίσιο αυτά που θα κάνουμε και ευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς συμβαδίζουν. Δεν μπορούμε να είμαστε επιτυχεί διεθνώς παγκοσμίως αν δεν είμαστε συνεκτικοί εντό της Ένωσης και αν δεν εφαρμόσουμε εδώ την κοινοτική προσέγγιση. Γιατί τα παραθυράκια θα παραμείνουν. Όλες οι πολιτικές μας πρέπει να στοχεύσουν ωστόσο πρωτίστως στην απασχόληση. Να δώσουμε δηλαδή την ευκαιρία στη νέα γενιά να βρει δουλειά βρίσκω επίσης ότι υπάρχει μια νέα όθηση, θα τα συζητήσουμε αυτά και στο θερινό συμβούλιο και χαίρομαι που ο πρόεδρος του έχει βάλει το θέμα αυτό τόσο υψηλά στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει να καλυφθούν τα κενά εκεί που έχουμε και να προχωρήσουμε και στην πράσινη οικονομία όπου υπάρχει ανάγκη να γίνουν επενδύσεις σε δεξιότητες που θα ακολουθήσουν την εξέλιξη αυτή. Οι αγορές εργασίας στην Ένωση και στο επίπεδο των κρατών και στο επίπεδο της Ένωσης πρέπει να είναι καταλήτης, όχι εμπόδιο για την πρόθεση του θέματος αυτού. Πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε τους υφιστάμενους πόρους και όλα τα δημοσιονομικά εργαλεία που διαθέτουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους στο εθνικό επίπεδο όπου μπορούμε. Πρέπει να στηρίξουμε δε τις πολιτικές μας αυτές με δάνεια προς τις επιχειρήσεις Προ του εργαζόμενου κτλ. ώστε να ανθίσουν καινούργιε δουλειέ για να μπει ο κόσμο στην αγορά εργασία. Που αυτό για μας είναι κέριο για να υπάρξει ανάπτυξη. Τα τελευταία δύο χρόνια η Ευρωπαϊκή Κομισιόν έχει βάλει ω πρώτη προτεραιότητα την καταπολέμηση τη ανεργία με όλες αυτές τις flagship initiatives που έχουν ε, προωθήσει ε, την προσπάθεια αυτή. Πρόσφατα η Κομισιόν ενέκρινε στις 5 Δεκεμβρίου του 2012 δηλαδή το πακέτο για την απασχόληση των νέων. Με μια εγγύηση που θα δώσει σε όλους τους νέους από 18-24 ετών τη δυνατότητα να συνεχίσουν είτε την εκπαίδευσή τους ή να μπουν σε μια ε, πρακτική εξάσκηση. Αντέδρασε ταχαίως η Επιτροπή για να υλοποιήσει την πρόταση αυτή επισημειώνοντας 6 δισεκατομμύρια ευρώ στο δημοσιονομικό πλαίσιο για να χρησιμοποιηθούν για τον σκόπο αυτό. Βέβαια αυτή η πρωτοβουλία ακόμα δεν έχει εγκριθεί και ανησυχεί η Κομισιόν βλέποντα ότι αποδυναμώνεται η φιλοδοξία των προτάσεών τη. Η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να προβλέψει και από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθεροποίηση αλλά και από όλα μία σημαντικά κονδύλια. Και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, από όπου προέκυψαν συγκεκριμένε συστάσει για τι χώρε μέλη, και θα τι δημοσιεύσουμε αυτέ αύριο, οφείλουμε να εξασφαλίσουμε ότι η ανεργία των νέων αντιμετωπίζεται σωστά και της δίνεται η σωστή προτεραιότητα. Στρατηγικές για την απασχόληση των νέων είναι κέριο σημείο, κέριο ε, στοιχείο για την ανάπτυξη. Ο χρόνος πιέζει όλες και όλους μας για να εφαρμόσουμε τις προτάσεις αυτές πραγματικά, να τις υλοποιήσουμε. Οι πολίτες μας έχουν θεμητές προσδοκίες από τους ηγέτες και από τα όργανα που πρέπει να κάνουν κάθε τι το δυνατόν για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν όλοι να συνεχίσουμε και μάλιστα να επιταχύνουμε το ρυθμό των προσπαθειών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία ε, σε αυτές τις συνεδριάσεις ακολουθούν οι ομιλητές ε, πέντε κύριοι και τρεις κυρίες που εκπροσωπούν τις πολιτικές τους ομάδες. Είναι ένα είδος κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ομάδας τους. Πρώτος ο κύριος Παόλο Ρανζέλ, εξ ονόματος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για 8,5 λεπτά παρακαλώ. Euh, Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου και τη Κομισιόν, αγαπητοί συνάδελφοι, την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδρίασε για να μιλήσει για την φοροδιαφυγή. Είναι ένα αναπόφευκτο θέμα, διότι ετησίω η Ευρώπη χάνει ένα τρει ευρώ, πάνω από ένα τρει ευρώ. Σε σύγκριση με τι ετήσιε δαπάνε μα για την υγεία, την παιδεία, την ασφάλεια, αυτό το νούμερο είναι εντυπωσιακό. Ορισμένοι μάλιστα παρατηρούν την απουσία αποτελεσμάτων μετά από την σύνοδο του περασμένης εβδομάδας. Θεωρούν πως ε, τα λόγια υπερίσχυσαν των πράξεων και πάλι δεν έχουν ακόμα απόλυτα άδικο. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι αυτά αποτελέσματα και αυτά τα αποτελέσματα μπορούμε να επιτύχουμε από κοινού με μια πραγματική ευρωπαϊκή ηγεσία. Ας μιλήσουμε τώρα για τους φορολογικούς παραδείσους. Ολόκληρο τον κόσμο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Ομισκοτικού Ταμείου, η φορολογική παράδοση είναι ε, της τάξης των 14-3 εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος αυτών συγκεντρώνεται στην Ευρώπη και αν δεν είναι άμεσα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο βρίσκονται σε ευρωπαϊκά προτεκτοράτα. Τίθεται λοιπόν θέμα ασυνέπειας εδώ. Φανταστείτε μία στιγμή μόνο. Αν κάθε χρόνο μπορούσαμε να συλλέξουμε το 20%, 20% από αυτό το έλλειμμα πόσο πολύ θα μπορούσαμε να μειώσουμε, μειώσουμε τα χρέη μας και πόσο θα μπορούσαμε να οθήσουμε τις ευρωπαϊκές επενδύσεις. Διαπραγματευόμαστε για την τελευταία δεκάρα για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο σε μια φάση όπου χρειαζόμαστε οπωσδήποτε την ανάκαμψη. Γι' αυτό και χρειάζεται ένα αυτόματο μήνυμα ενημέρωσης να φτιαχτεί ανάμεσα στις ε, φορολογικέ αρχές των κρατών μελών. Επίσης είναι ε, απαραίτητο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ε, περί αποταμιεύσεων. Πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί με τους φορολογικούς παραδείσους. Και υπάρχει ένα ακόμα σημείο που με ενοχλεί. Είναι η κατανομή της αναπτυξιακής βοήθειας σε χώρες οι οποίες ταυτόχρονα έχουν ε, και δέχονται ευρωπαϊκά κρυφά ευρωπαϊκά ενεργητικά και που μαζί με τους ευρωπαϊκούς φορολογικούς παραδείσους ωφελούνται από τις ευρωπαϊκές υποδομές της ενιαίας αγοράς, της ασφάλειας, των κοινών μας πολιτικών και σε αντάλλαγμα κρύβουν χρήματα που ακριβώς θα έπρεπε να ενισχύουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Στα γαλλικά αυτό το λένε ότι θέλουν και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Ε, αλλά αν θέλουμε εμείς πραγματικά να είμαστε λογικοί, οφείλουμε να φτάσουμε στο τέλος αυτού του συλλογισμού. Έχουμε υπερασπιστεί εντόνως το διπλό πακέτο και το εξαπλό πακέτο μέτρων. Την περασμένη εβδομάδα υπερψηφίσαμε τον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας. Και όλα αυτά τα κάναμε για να έχουμε μια αποτελεσματική οικονομική ένωση που θα είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να μπορεί να αποφύγει μελλοντικά ε, σοκ. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο, διότι όλα αυτά δεν θα είναι αποτελεσματικά παρά μόνο αν έχουμε αντιμετωπίσει σαφώς το θέμα της ευρωπαϊκής φορολογίας. Ε, για να βγούμε από την κρίση δεν αρκεί να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή, και η φορολογική παράδειση πρέπει να γίνουν ε, σταθερά βήματα προς ένα ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα. Ένα σύστημα που θα είναι μόνο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Γιατί διαφορετικά τι θα γίνει, θα επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα που κάναμε με την ενιαία αγορά. αφήνοντας 150 σημεία παγωμένα που θα έπρεπε να έχουν ρυθμιστεί από το 1992. Αποτέλεσμα, 20 χρόνια μετά, ακόμα για τα ίδια μιλάμε. Οι πολίτες μας χαίρουν ελευθεριών τις οποίες εγκιάται η Ευρώπη, αλλά από τη στιγμή που γίνεται λόγος για φορολογία, είναι λες και η συνθήκη της Ρώμης δεν είχε ποτέ υπογραφεί. Χρειάζεται μεγαλύτερη σύγκληση στα οικονομικά και κοινωνικά μας πρότυπα βεβαίω, αλλά χρειάζεται επίσης και μεγαλύτερο φορολογικό συντονισμό, αν όχι και φορολογική εναρμόνιση προ μια πραγματική δημοσιονομική, τραπεζική και φορολογική ένωση. Αντί γι' αυτό όμως, κάθε χώρα έχει διαφορετική φορολογική στρατηγική Άλλε φορές φορολογείται η αποταμίευση, άλλε φορές η ακίνητη περιουσία, άλλε άλλες φορές ε, η μισθή και έτσι χάνουμε χρόνο και χρήμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλησα να μιλήσω στα γαλλικά μέχρι τώρα, γιατί αντιπροσωπεύω τον πρόεδρο Ζωζεφ Ντόλ. Τώρα επιτρέψατε μου να χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα, διότι θα επιθυμούσα να σας μιλήσω για τις ε, χώρες ε, που δέχονται οικονομική βοήθεια όπως η χώρα με η Πορτογαλία. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω πως κατέστη σαφέ πως ε, το ΕΛΚ ε, σε σχέση, ε, υπογραμμίζει τις πρόοδους που σημειώθηκαν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά είναι ακόμα απόρο απέχουν από αυτά που επιθυμούσαμε. Η ευρωπαϊκή οικοδόμηση απαιτεί την οικοδόμηση μιας τραπεζική, δημοσιονομικής και φορολογικής ένωσης δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους μόνο, παρά μόνο αν έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία και πραγματική φορολογική εναρμόνιση που θα επιτρέψει να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση και Οικονομική Ένωση η οποία ε, και δεν θα κατακαιρματιστεί. Ε, έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια ομοιογένεια φορολογική στην Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη, πράγμα που δεν εμποδίζει ούτε θα πρέπει να εμποδίσει τη δημιουργία φορολογικών κινήτρων είτε ζώνε σε θετικής φορολογικής ε, Από τη στιγμή που ισχύει αυτή η φορολογική διαφορά, διαφορά χωρίς λογική, χωρίς διαφάνεια και χωρί συγκεκριμένα και καθολικά κριτήρια, και μιλώντα ε, για τι χώρε που αντιμετωπίζουν τι μεγαλύτερε δυσκολίε και που δέχονται οικονομική βοήθεια όπω η δική μου χώρα η Πορτογαλία εδώ υποστηρίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει απορρίθμιση φορολογική σε σχέση με ε, το φόρο επί των επιχειρήσεων ω προκίνητρο για τι ε, επιχειρήσει ω ένα κίνητρο για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Η φορολογική εναρμόνιση, η φορολογική συνέπεια και συνοχή δεν σημαίνει ενιαίο και καθολικό και ομοιόμορφο πλαίσιο για ολόκληρη την Ένωση. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι οι πιο πλούσιε χώρες έχουν πολλές φορές πιο ευνοϊκή φορολόγηση, ενώ εκείνε που χρειάζονται επενδύσεις και ανάπτυξη που αντιμετωπίζουν τεράστιε δυσκολίες έχουν πολύ μεγάλη επίση δυσκολία στο να εγκρίνουν φορολογικά καθεστώτα που να δίνουν κίνητρα. Χρειαζόμαστε συνεπέ πλαίσιο όπου τα έσοδα και δεν θα είναι στην υπηρεσία κάποιων χωρών που πολύ συχνά είναι και πιο ανταγωνιστικές της Ένωσης, αλλά που θα χρησιμοποιούνται ως μέσα πολιτικής ε, οικονομικής για να ε, μπορέσει να ανακτηθεί και να αποκατασταθεί η οικονομία η πιο ε, ζημιωμένη στο πλαίσιο της Ένωσης. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν όλες οι διαφορές, αλλά ότι θα υπάρξει ορθολογισμός, διαφάνεια, ε, και συγκεκριμένα κριτήρια. Με λίγα λόγια, εάν ε, υπάρξει συνοχή, συνέπεια και διαφάνεια στα φορολογικά συστήματα των χωρών της Ένωσης, είμαστε πεπισμένοι ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε στις χώρες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες ένα φορολογικό σύστημα προσαρμόσιμο που θα μπορέσει να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα ελλείμματα και οι δυσκολίες. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της Επιτροπής και τον πρόεδρο του Συμβουλίου κάνω μια έκκληση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να ενθαρρύνουν και να δεχτούν μέσα σε αυτό το πνεύμα μια φιλόδοξη φορολογική μεταρρύθμιση του καθεστώτος φόρου των επιχειρήσεων στις χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό συγκεκριμένα προγράμματα και συγκεκριμένα για τη χώρα μου την Πορτογαλία. Νομίζω ότι μόνο καταπολεμώντα τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή, του φορολογικού παραδείσους, μέσω τη εφορολογικής εναρμόνισης θα έχουμε αρκετό χώρο για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα όπου η πρόσβαση στις εξαιρέσεις θα είναι στην υπηρεσία των πιο φτωχών ε, ε, και, των λιγότερο ευνεμένων περιοχών και όχι στην υπηρεσία των πιο ανταγωνιστικών περιοχών και ζωνών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Παύλο θα παρακαλέσω όλους τους συναδέλφους να προσπαθούν να τηρούν το χρόνο τους για να ε, τελειώσουμε εντός του πλαισίου. Εμείς οι σοσιαλιστές συνήθως είμαστε πάρα πολύ ε, μακρόθυμοι με τους χριστιανούς συναδέλφους, αλλά δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύεστε αυτή την καλοσύνη μας, παρακαλώ. Ο κύριος Βόμποτα έχει το λόγο, εξ ονόματος ε, των δημοκρατών και σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ λέει ο κύριος Φόβοδα. Σήμερα ήρθε στα λόγια μας ο κύριος Ρανζέλ. εμεί τα έχουμε πει αυτά εδώ και δύο-τρία χρόνια. Αυτή είναι η πρόοδος. Ε, ε, καταλαβαίνουν σιγά-σιγά αυτά που λέγαμε εμείς εδώ και τόσα χρόνια. Είπατε κύριε Ρομπαϊ ότι ήταν μικρή, σύντομη συνεδρίαση, πλην όμως αποτελεσματική. Ίσως αυτό να πρέπει να γίνεται ε, σύντομη συνεδρίαση, αλλά με την ενεργειακή απόδοση ποτέ δεν μπορεί να είσαι αρκετά αποδοτικός, ούτε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να εξηγήσω γιατί. Για την ενέργεια. Εδώ και χρόνια, όχι μόνο εμείς, ε, εργαζόμαστε για μια ενεργειακή κοινότητα. Συγγεί χθείως στο Συμβούλιο και τα μέλη του. Τώρα το προχωρούν. Ωραία, επιτέλους, το κατάλαβαν. Εδώ και χρόνια εμείς αγωνιζόμαστε για μια κοινή αγορά ενέργειας. Δύο-τρία χρόνια τώρα έρχονται και εκείνοι στα λόγια μας. Μια μεγάλη χαλιβουργική ε, στην πόλη μου, στο Λίντς, ε, μας εξήγησε για ποιο λόγο ε, οι νέε εταιρείε θα μετακατασταθούν στις Ηνωμένε Πολιτείε αν του επιτραπεί ε, ο νέος τρόπος λειτουργίας. Ε, για ποιο λόγο, όχι επειδή υπάρχει άλλο πρόβλημα κοινωνικό, μισολογικό στην Ευρώπη, αλλά το κόστος της ενέργειας είναι το μισό στις Ηνωμένε Πολιτείε είμαστε ε, πολύ ε, θαραλέοι για την υδρορογμάτωση, αλλά για τα υπόλοιπα θέματα οι Ευρωπαίοι δεν προχωρούμε αρκετά. Και πραγματικά υπάρχουν τεχνολογίες σοβαρές και ε, ασφαλείς για το περιβάλλον. Αυτό που μας χρειάζεται είναι ενεργειακή απόδοση και πάλι το γνωρίζετε και εσείς κύριε Βαρόσο, ξέρει πόσο, πόσοι μήνες χρειάστηκαν, τα ξέρουν εδώ οι παρευρισκόμενοι, για ένα στόχο δεσμευτικό και τελικά δεχτήκαμε ένα συμβασμό, Διότι ε, οι διακηρύξεις είναι κάτι καλό, αλλά οι πράξεις είναι κάτι διαφορετικό. Φόρο διαφυγή. Εξηγήσατε κύριε Βαρόπε και το σημείωσα ότι οι διαπραγματεύσεις με Ελβετία, Λιχτεστάιν και λοιπά θα γίνει βάση της αναθεωρημένης οδηγίας για τη φορολόγηση των καταθέσεων. δεν το κατάλαβε κανείς αυτό ούτε στο Λουξεμβούργο ούτε στην Αυστρία. Εμείς είχαμε καταλάβει πρώτα να διαπραγματευτούμε και μετά ε, θα δούμε. Όχι, ε, εγώ ε, σημειώνω αυτά που είπατε και τα παίρνω σοβαρά βάση της αναθεωρημένης οδηγίας. Και τα δύο χρειαζόμαστε, αλλά και πολύ περισσότερα. Το είπε και ο πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα το αναλύσουν και άλλοι συνάδελφοι. Ε, θα πρέπει να κλείσει η φορολογική ψαλίδα μέχρι το 2020, να δούμε τι κάνουν οι πολυεθνικές. Αυτό συζητούν και η Apple και οι άλλοι. Πολλές πολυεθνικές εκμεταλλεύονται ε, για να φοροδιαφεύγουν τα διάφορα φορολογικά συστήματα και να πληρώνουν πάρα πολύ χαμηλούς φόρους. Ε, είναι κάτι που αφορά και άλλες εταιρείες και ιδιαίτερα τις τράπεζες. Ε, έρχομαι τώρα, μου επιτρέπετε, σε ένα τελευταίο στοιχείο, πολύ σημαντικό για μας, και αυτό είναι η ανεργία των νέων. Χάρηκα πάρα πολύ κύριε Βαν που αναφερθήκατε στο θέμα αυτό. Διότι τι βλέπουμε αυτό τον καιρό. Και πάλι συμφωνώ με τον κύριο Μπαρόζα από αυτού και ελπίζω και εσείς να συμφωνείτε. Τι βλέπουμε αυτό τον καιρό. Βεβιασμένες κινήσεις, ξαφνικά. Τόσα χρόνια ανέβαινε η ενέργεια των νέων, τώρα αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι. Τώρα όλοι τρέχουν στην Ισπανία, στην Ελλάδα και αλλού για να τους βοηθήσουμε. Γερμανός υπουργό και η γερμανική κυβέρνηση βοηθάει, βεβαίως. Βοηθάει. Πέντε 5.000 ε, από 3 εκατομμύρια νέους θα έχουν κάποια εκπαίδευση. Ε, κάτω των 35 ετών. Εντάξει, είναι θετικό. Επιτέλους, κάτι κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το αφήνουμε αυτό σε μεμονωμένες κυβερνήσεις που ξαφνικά διαπιστώνουν ότι είναι χριστιανοί φιλάνθρωποι και να βοηθήσουμε τους φουκαριάριδες αυτούς τους νέους ανέργους. Πρέπει να είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Ωραίε είναι οι διακηρύξει, αλλά η δράση που είναι και ο προπολογισμό. 6 δισεκατομμύρια για όλε τι χώρε, όχι όλε, τι περισσότερε. Για μία επταετία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σταγόνα στον ωκεανό. Μπορεί να είναι σημαντικό για ορισμένους μεμονωμένα, αλλά δεν θα σωθεί η Ευρώπη έτσι. Γι' αυτό ζητούμε και αυτό τον οπισθοβαρή προγραμματισμό στον προπολογισμό, το backloading. Αλλά όχι σε σχέση με το τι θα γίνει μετά, αλλά να έχουμε βρει τα χρήματα και τα ευρώ να υποστηρίξουμε και την εγγύηση για την νεολαία και τις επόμενες χρονιές. Διότι δεν θα σταματήσει ξαφνικά, δεν θα εξαφανιστεί η ενεργεία των νέων το 2015 τέρμα ή το 2016. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Και ο Γερμανός Υπουργός και ε, συναντήθηκε και με τον Γάλλο Υπουργό και ο δικό μου υπουργό έχει πάει στην Ισπανία, δεν με. Καλό είναι να αυξάνεται η συνειδητοποίηση του μεγέθου του προβλήματο, αλλά χρειαζόμαστε μια γνήσια ευρωπαϊκή πολιτική. Εσεί αποφασίσατε για την εγγύηση στην νεολαία μετά την πρόταση τη Κομισιόν και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μέχρι σήμερα τι έγινε. Πριν από ένα χρόνο αποφασίσατε για το Σύμφωνο ανάπτυξη και μέχρι τώρα τι έχει γίνει θέλω να δραστηριοποιηθείτε εσείς περισσότερο και να ζητήσετε από τους συναδέλφους σας στις κυβερνήσεις πραγματικά να δράσουν. Ωραία τα λόγια, χρειάζονται και έργα στην Ευρώπη όμως. Και εσείς και εμείς οι βουλευτές θα κατεβούμε στις εκλογές αύριο. Τελειώνει η παρούσα θητεία, η θητεία και για σας. Πώς θα βγούμε στους νέους να πούμε κάναμε κάτι για σας, αγωνιστήκαμε κατά της ε, ανεργία των νέων. Αγωνιστήκαμε για να έχετε μέλλον στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι για μας η μεγάλη πρόκληση και ελπίζω πραγματικά εκεί να δοκιμαστούμε στην πραγματικότητα. Οι νέοι δηλαδή να έχουν μια ευκαιρία να βρουν επιτέλους δουλειά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Χάνες. Εξ ονόματος των Δημοκρατών και Φιλελευθέρων τώρα για τρία λεπτά η κυρία Βαλεάν παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Κύριε Πρόεδρε Βαν Ρόμποϊ, δώσατε την εντύπωση ότι και το Συμβούλιο κατανοεί ότι αποτυχαίνει η Ευρώπη. Όχι μόνο οι ενεργειακές μας τιμές είναι τριπλάσιες των ΗΠΑ της Αμερικής. Μάλιστα και παρά τις, τις ε, πολιτικές μας για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, παρόλα αυτό τα καυσαέρια αυξάνονται. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Η δική μου πολιτική ομάδα των φιλελευθέρων θεωρεί ότι ο μόνος τρόπος να αναστραφεί η τάση αυτή είναι να ξεκαθαριστεί η κατάσταση της αγοράς σε ό,τι αφορά τους επενδυτές. Όσο οι επενδυτές δεν γνωρίζουν ποιο θα είναι το μελλοντικό νομοθετικό πλαίσιο, θα παραμείνουν διστακτικοί. Δεν θα επενδύουν ούτε σε ενεργειακά δίκτυα, ούτε σε αποδοτικότητα της ενέργειας, ούτε στην ε, αντιμετώπιση ούτε στην πρόθεση των ανανεώσιμων ενεργειών. Τα λέμε αυτά εδώ και πολύ καιρό. Μιλούμε τώρα για το φυσικό αέριο, για νέες τεχνολογίες. Λέτε εσείς ότι θα τα περιλάβετε στις πολιτικές σας. Πρέπει να είστε σαφέστεροι και όχι απλώς να υπονοείτε. Το Συμβούλιο στο, στη συνάντησή του νομίζω μάλλον ότι το, ε, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ήταν μια μεγάλη ευκαιρία που νομίζω ότι χάθηκε και δεν θα υπάρξουν αλλαγέ πολιτική στι χώρε μέλη. Θέλω να τονίσω λοιπόν εδώ τρία πράγματα. Πρώτο, την εφαρμογή του τρίτου πακέτου τη ενέργεια. Αυτό είναι προτεραιότητα. Είναι κάπω αργά ήδη βέβαια, για να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Είπατε κι εσεί κύριε Μπαρόσο ότι ήταν ένα μεγάλο θέμα και τη προηγούμενη θητεία σα το πακέτο της κλιματικής αλλαγής, το πακέτο της ενέργειας και ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί και δεν περπατάει το σύστημα της ε, εμπορίας των ε, εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, το ETS. Εδώ λοιπόν πρέπει να σημειωθεί δράση. Η ενιαία ενεργειακή αγορά εξακολουθεί να απέχει από την πραγματικότητα για λόγους ότι ακόμα δεν έχουν μεταφέρει στις, ε, στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις του πακέτου ορισμένες χώρες μέλη, μεγάλες μάλιστα χώρες μέλη, και επομένω εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια στη δημιουργία τη ενιαία αγορά. Ε, Δεύτερον, συμφωνούμε με το συμπέρασμά σα ότι οι επενδύσει σε ε, ε, καινοτόμα δίκτυα ανανεώσιμων ενεργειών είναι απαραίτητε. Όμω, δεν συμφωνούμε απόλυτα με τη δράση που αναλαμβάνει το Συμβούλιο για υπέρ τη διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη, όπου εγώ είμαι εισηγήτρια και γνωρίζουμε καλά, πρώτον από 9,9 δισεκατομμύρια που πρότεινε η Κομισιόν, τα έκοψε σε, στα μισά, 4,51 το Συμβούλιο. Δεύτερο, υποτίθεται ότι θα λαμβάνονταν 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα όμως περικόπτει όπως είπα το Συμβούλιο, της δαπάνες. Δεν θα είναι δυνατόν με τα μικρά αυτά ποσά να χρηματοδοτήσει τι προτεραιότητες που περιλαμβάνετε στην περάσματά σας. Σας ζητούμε λοιπόν να επανεξετάσετε την θέση σας σχετικά με τη δημοσιονομική προκοδότηση του ε, έργου συνδέοντα στην Ευρώπη. Έχουμε τώρα και στην ασυνέχεια μεταξύ των συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των πολιτικών που ακολουθεί. Εσείς συμπεραίνετε ότι η επένδυση για τις υποδομές ενέργειας θα προέλθουν από την αγορά. Εδώ σας στηρίζουμε απολύτως εμείς οι φιλελεύθεροι. Ωστόσο, αν το πιστέψουμε αυτό, τότε, αν πιστέψουμε δηλαδή ότι η χρηματοδότηση θα προέλθει από την αγορά, πρέπει να υποστηρίξετε τότε τα εργαλεία εκείνα τα οποία θα αντλήσουν τα απαραίτητα κονδύλια από την αγορά. Εκεί χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Συμβουλίου για τα ομόλογα έργων και για τα άλλα σχετικά δημοσιονομικά ε, ή χρηματοδοτικά καλύτερα εργαλεία. Ευχαριστώ εξ ονόματος των Πρασίνων για τρία λεπτά επίσης η κυρία Χάμς. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Στο τελευταίο Συμβούλιο πράγματι έγιναν κάποιες κινήσεις γύρω από το θέμα της φορολογίας, έτσι το εκτιμά η ομάδα μου ότι δηλαδή το τραπεζικό απόρριτο αρχίζει να σπάει και ότι επομένως ελπίζω, ελπίζω μακάρι η φοροδιαφυγή, η παράνομη φοροδιαφυγή να μπορέσει να αντιμετωπιστεί στο μέλλον. Αυτό που βλέπουμε εμεί ωστόσο κριτικά είναι ότι το Συμβούλιο δεν μπόρεσε ξανά να προτείνει και να αποφασίσει πέτρα που θα οδηγήσουν ώστε οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις να μην μπορούν να αποφεύγουν τις φορολογικές υποχρώσεις στις χώρες όπου αποκομίζουν τα κέρδη τους. Εξακολουθεί να παραμένει αυτό ένα μέγα ανοιχτό κεφάλαιο. Πρόκειται για φορολογικό dumping. Ένας άγριος ανταγωνισμός εδώ στην Ευρώπη για τα φορολογικά που δεν έχει σταματήσει. Και κύριε Βαν Ρόμποϊ, τι εννοούσατε όταν είπατε ότι η προθεσμία για την διευκρίνηση όλων των ανοιχτών θεμάτων θα είναι το Δεκέμβριο φέτος. Εγώ κατάλαβα ότι εκεί θα αποδώσετε λόγο και ότι τα θέματα, τα ανοιχτά θέματα θα τεθούν. Deadline για απόφαση, εγώ δεν βρήκα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Εν προκειμένου με ενδιαφέρει πολύ ποια είναι η θέση σας ως Συμβούλιο σχετικά με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την αναχώρα προσέγγιση δηλαδή που είχε βρει αρχικά θετική απήχηση στο Συμβούλιο, πώς μπορεί λοιπόν αυτό να επανέλθει η Επιτροπή μας, η, οικονομική, η ΕΚΟΝ, είχε προτείνει και η Sharon Bowles, η πρόεδρός της, είχε προτείνει οδηγίες για τη διαφάνεια, οδηγία για τα ε, λογιστικά πρότυπα. Εκεί πρέπει να συνεννοηθούν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Τώρα, δεύτερο, ενέργεια. Μιλήσατε για επανάσταση της ενέργειας. Δυστυχώς εδώ οφείλω πάλι να είμαι σκληρή μαζί σας. Εγώ νομίζω ότι εδώ αυτό που κάνετε είναι αντεπανάσταση. Κάθε τι, το λογικό, με το οποίο είχε ξεκινήσει ο Επίτροπος Άντρες Πίμπαρξ στην προηγούμενη θητεία για μελλοντικέ για στρατηγικές δηλαδή που είχαν κάποιο μέλλον, καθώς επίσης και με τον Επίτροπο Δήμα που είχαν αρχίσει κάποια πράγματα για μια πολιτική αντιμετώπιση των αλλαγών του κλίματος, όλα αυτά καταραίουν Εγώ βρίσκω παράλογο να μιλείτε για επιδοτήσεις νέων ατομικών εργοστασίων. 50 χρόνια μετά από την εισαγωγή του στην αγορά να μιλείτε τώρα πάλι για εισαγωγή στην αγορά. Και βρίσκω ακόμα πιο παράλογο την ιδέα ότι όσο πιο φτηνό θα είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, τόσο καλύτερα θα λειτουργήσει η οικονομία. Επομένω, θα προκύψει ξανά ε, οικονομική ανάπτυξη. Το ε, πετρέλαιο που βγαίνει από το σχιστόλιθο ίσω βράχει πρόθεσμα, αλλά για λίγο χρονικό διάστημα να επιτρέψει κάποια ε, ανάκαμψη. Αλλά νομίζω ότι πάει να ξεκινήσει εδώ μια ολόκληρη φούσκα η οποία θα σκάσει και θα έχει βαρύτατες επιπτώσεις. Τρίτο θέμα που θέλω να θίξω, που είναι το θλιβερότερο από όλα και αυτό δεν αφορά τόσο πολύ τις αποφάσεις του, του, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, περισσότερο τις αποφάσεις των υπουργών εξωτερικών. Η αντίληψη που έχω εγώ για, την εξελίξη, για τις εξελίξεις στη Συρία είναι πολύ σκοτεινή. Δεν μίλησαμε ακόμα γι' αυτό στην ομάδα μου. Αλλά έχω την εντύπωση ότι αν τώρα πραγματικά μετά τον Αύγουστο η Μεγάλη Βρετανία και η Αγγλία ως δύο μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας μαζί με τη Ρωσία που επίσης είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας από τα συνολικά πέντε προχωρήσουν σε εξοπλισμό, σε ανταγωνισμό εξοπλισμών στη Συρία προχωρούμε τότε σε ένα πόλεμο στη Συρία με, με πληρεξουσίους Κάτι εξουσιοδότηση Εάν σταματήσει δηλαδή μετά τον Αύγουστο το εμπάργκο. Ελπίζω να αποφευθεί αυτό το σενάριο. Θα ήθελα πολύ η κυρία Άστον και οι Υπουργοί Εξωτερικών να αναλάβουν αμέσως δράση για να μην υλοποιηθεί το σενάριο αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χάρμς. Για να είμαι ειλικρινής, καμιά φορά με επικρίνουν ότι κόβω τους ομιλητές στο μέσο της φράσης. Το πρόβλημα με τα γερμανικά είναι ότι δεν ξέρεις πού είναι το μέσο της φράσης, γιατί το ρήμα έρχεται στο τέλος, γιατί τραβάτε την πρώτη, τραβάτε, τραβάτε για να μην μπορώ να σας κόψω. Λοιπόν, για τρία λεπτά και πάλι θα δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Κάλαναν που θα μιλήσει εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Παρακαλώ. Even though we don't have our verbs at the end of the sentence, Ακόμα και αν ε, το δικό μας ζευρήμα δεν έρχεται στο τέλος ε, της φράσης, ελπίζω ότι δεν θα με κόψετε, αγαπητέ Ισπανέ συνάδελφε. Μια ένα πρόσφατο δημοψήφισμα στη δική μου περιφέρεια δείχνει ότι η πρώτη ανησυχία του κόσμου είναι αυτή τη στιγμή ψηλές τιμές της ενέργειας Και φαντάζομαι και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιφέρειες το ίδιο θα δείξει ένα δημοψήφισμα. Από το 2005 το κόστος ε, του ηλεκτρισμού έχει αυξηθεί κατά 1% στην Ιαπωνία, κατά 5% στη ΣΥΠΑ, στην Ένωση κατά 29% και στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 18%, 80% με συγχωρείτε. Ωστόσο, καλωσορίζουμε την απόφαση να εστιαστεί το πολιτικό κεφάλαιο σε αυτό το τομέα και οι προτεραιότητε που εξέθεσε το Συμβούλιο, δηλαδή επάρκεια στην ενέργεια, ενιαία αγορά, επενδύσει και διαφοροποίηση πηγών, μπορούν να επιτευχθούν μέσω ευέλικτη νομοθεσία που θα δώσει κίνητρα στα κοινικοκυριά και στι βιομηχανίε για να επιδιώξουν αυτέ τι πολιτικέ και όχι, ελπίζω, μέσω αυθαιρέτων στόχων και μέσω ομοιόμορφων μέτρων για όλους. Ούτως ή άλλως οι αυθαίρετοι στόχοι που εφευρέθηκαν για να ταιριάξουν στα ανακοινοθέντα τύπου, ενώ οι τιμές ε, της ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη οδηγούν ε, στο να κλείνουν τα εργοστάσια πριν να έχουμε αντικατάσταση, υποκατάστατα μάλλον ε, στις ενεργειακές πηγές. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα, δεν θα γίνουν ε, ούτε καν μετά που θα έχει φύγει ο κύριος Βαν Ρόμποϊ από αυτή τη θέση. Ελπίζω πως δεν θα, δεν θα μείνουμε από ενέργεια, δεν ξεμείνουμε στο μέλλον. Τώρα, ε, από ό,τι φαίνεται στο Συμβούλιο, ε, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι θέλαν να μιλήσουν για το λάδι, όχι το πετρέλαιο, αλλά το λάδι, το ελαιόλαδο και οι περισσότεροι πολιτικοί αποδεικνύουν ότι κάνουν λάθος ε, και πολλοί από εμάς προσπαθήσαμε να αποθαρρύνουμε τον Ντανιέλ ε, Κονπεντίτ από αυτή την ε, θεώρηση. Ωστόσο καλωθορίζουμε το είναι θέση του Επιτρόπου Τσιόλος. Δεν είναι βέβαια το τέλος της προσπάθειας. Δείχνει ωστόσο ότι πιστεύουμε πως οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν ε, δεν τους εμπιστευόμαστε ούτε καν για να αποφασίσουν πώς θα καταναλώσουν το λάδι στα εστιατόρια. Ελπίζω πως αυτή η απαγόρευση τελικά θα ε, ξεπεραστεί σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, είπα την περασμένη εβδομάδα ότι η συνεργασία για να παρεμποδιστεί η παράνομη φοροδιαφυγή θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγκάλυψη για να περάσει εναρμόνιση όλων των ε, φόρων, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως μια εναρμόνιση δεν θα είναι προς τα κάτω. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά ανταγωνιστική παγκοσμίω, χωρίς να κάνουμε την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Και γι' αυτό ναι, ανησύχησαν ιδιαίτερα οι παρατηρήσει του Προέδρου Σούλτ μετά από το Συμβούλιο την περασμένη εβδομάδα όταν είπε ότι έχουμε ανταγωνισμό φορολογικό εντό τη Ένωση, πράγμα το οποίο δεν είναι πολύ λογικό. Γι' αυτό ελάχιστε προδιαγραφέ υπό ότι στο πλαίσιο των φορών θα πρέπει να ισχύσουν και νομίζω και ότι ο Επίτροπος έμετα θα προτίθεται να κάνει μια βασική πρόταση γι' αυτά. Ελπίζω να έκανε λάθος, ελπίζω να είναι λάθος ε, τα όσα μου είπαν και ελπίζω κύριε Πρόεδρε πως δεν θα αναζητήσει την εναρμόνιση της φορολογία με τέτοιο τρόπο ώστε να λήξουν τα διανταγωνιστικά φορολογικά ποσοστά τα οποία βοήθησαν χώρες όπως η Ιρλανδία να ξεπεράσουν την ε, κρίση, την ύφεση. Ε, ακόμα και η εισαγωγή μήνυμου με επίπεδα θα ήταν μέγα σφάλμα πολιτικός και οικονομικός. Αν οι χώρες θέλουν να εισάγουν ε, μη ανταγωνιστικά φορολογικά ποσοστά, δημοκρατία έχουμε, είναι το δικαίωμα του καθενός, αλλά να μην τραβήξουμε όλους ε, στα επίπεδα της Γαλλίας έτσι ώστε ο Λάντα απλώς να φαίνεται λιγότερο καταστροφικός στην πολιτική του. Ε, Ευχαριστώ κύριε Καλανάν. Εξ ονόματο της ομάδας Ελευθερία και Δημοκρατία, το λόγο έχει ο κύριο Περόνι για δύο λεπτά. Κανονικά θα έπρεπε να λάβει το λόγο για δυόμιση λεπτά, είπαμε. Σας ευχαριστώ. Η Κομισιόν περισσότερο παρατηρήσεις έκανε και όχι συγκεκριμένες αποφάσεις. Δεν έλαβε συγκεκριμένες αποφάσεις. Θα δούμε πότε όλα αυτά και αν θα εφαρμοστούν ποτέ. Όσον αφορά όμως πραγματικά την Ένωση, αυτό που ενδιαφέρει είναι η συμμετοχή των πολιτών. Από το να αφήνουμε διαρκώς ε, την πίσω μας την ε, κοινή βούληση, ε, εκτός από τις μέρες των εκλογικών αναμετρήσεων, δεν μπορεί να οδηγήσει σε τίποτα το θετικό. Η απομάκρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά της όργανα, τα σημεία τα ισχυρά της, όπως το ευρώ, όπως ο χώρος Σέγγεν, αυτή η αδιαφορία και απομάκρυνση διαρκώς αυξάνεται. Ολισμένοι το θέλουν, άλλοι πολύ λιγότερο. Απάντως είναι γεγονός. Και με εκκλήσεις ή αποφάσεις ε, που λαμβάνονται κεντρικά και γραφειοκρατικά ε, δεν πρόκειται να επιτευχθεί μια νέα εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, θα έπρεπε να μπορέσουμε να κάνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν περισσότερο, έχοντας αυτό το θάρρος που μέχρι τώρα μας έχει λείψει και να τους θεωρούμε όχι υπηκόους, όχι παθητικούς υπηκόους, αλλά ε, υποβάλλοντας σε δημόσια δημοψηφίσματα, όπως κάνει η Ελβετία, που βέβαια τα καταφέρνει πολύ καλύτερα στην κρίση, ίσως ακριβώ επειδή δεν είναι στην Ένωση, ίσως επειδή δεν είναι στο ευρώ, ίσως επειδή έχει μια φορολογική πολιτική πολύ χαμηλή από, αυτές τις, από αυτή των χωρών της Ένωσης. Να υποβάλουμε λοιπόν σε δημοψηφίσματα τα φετίχ της Ένωσης, ε, ξεκινώντας από το ευρώ, για να έχουμε μια συνένεση ή μια απόρριψη από πλευράς όσων πραγματικά είναι οι εγγυητές της κυριαρχίας, δηλαδή τους λαούς. Αυτό που ζητούν η Λέγκα του Βορρά και άλλες συνιστώσεις της ομάδας που αντιπροσωπεύω είναι αυτό που ζητούν και οι πολίτες της Ευρώπης, της Ένωσης, για να υπάρξει μια πραγματική δημοκρατία. Gracias, señor Speroni. Ευχαριστώ κύριε Σπερώνη. Εξ ονόματος της Ενωτικής Αριστερά για 2,5 λεπτά η κυρία Τσίμερ παρακαλώ. Κύριε Μπαρόσο, είπατε προηγουμένως ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ε, η οι αποφάσεις που έλαβε το Συμβούλιο είναι στη σωστή κατεύθυνση και προφανώς αυτό εννοείται ότι είναι σωστά προσανατολισμένες. Εγώ το αμφισβητώ αυτό διότι βλέπω μια αλλαγή παραδείγματος στη διάρκεια των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και μάλιστα και στα συμπεράσματα του ήδη με την πρώτη φράση των συμπερασμάτων, εκεί όπου λέει δηλαδή ότι τώρα πια πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα και να επιτύχουμε την ανάπτυξη. Αυτά δεν είναι τυχαίες διατυπώσεις. Και μάλιστα Όλε οι αποφάσει υπάγονται του Συμβουλίου σε αυτό, αυτή την αλλαγή παραδείγματο. Επομένω, το μήνυμα είναι ότι στην ουσία πρόκειται για μια βάρβαρη περιθωριοποίηση όλων των απαιτήσεων περιβαλλοντικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών κοινωνικών και Όλα αυτά θα πούνε στην άκρη, εφόσον δηλαδή θα πρόκειται μονάχα για αγώνα υπέρ τη διεθνού ανταγωνιστικότητα. Το Συμβούλιο κανονικά έπρεπε να αντιμετωπίσει την πρόκληση να σταματήσει την οικολογική καταστροφή. Αλλά για παράδειγμα, αντί να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της, εν, της παινίας ενέργειας, δηλαδή άνθρωποι που δεν έχουν ούτε για να ζεσταθούν, τώρα πάει να μειώσει τις τιμές υπέρ της μεγάλης βιομηχανίας, επιβαρύνοντας παραπάνω τους καταναλωτές. 15 εκατομμύρια και παραπάνω άνθρωποι στην Ένωση δεν έχουν αρκετά λεφτά για να πληρώσουν το λίγο ρεύμα που χρειάζονται για να ζεσταθούν και για να μαγειρέψουν. Αυτά τους αρνείστε εσείς και αυτά που προβάλλεται ως δίθεν αποδοτικότητα στη χρήση της ενέργειας και ασφάλεια της προμήθειας πάνε σε μια κατεύθυνση που δεν προστατεύει τους ανθρώπους απέναντι στην αγωνία που έχουν ότι το γκάζι που θα χρειάζονται να, για να μαγειρέψουν, για να ζεσταθούν στην ουσία συνεπάγεται καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Το θέμα που θα πρέπει είναι ποιος παράγει, πώς και για ποιον ενέργεια. Από εκεί πρέπει να προκύψουν όλα τα υπόλοιπα και για παράδειγμα και η φορολόγηση της ενέργειας και μια προσπάθεια βιώσιμης παραγωγής και χρήσης της ενέργειας. Οι διατυπώσεις που επιλέχθηκαν τελικά βαίνουν στην απολύτως αντίθετη κατεύθυνση. Για παράδειγμα fracking, δηλαδή θράψη των σχιστολίθων για να εξαχθεί πετρέλαιο, υδρορογμάτωση ενώ θα έπρεπε να φροντίσετε να δώσετε ενέργεια στον κόσμο, στους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό θα σήμαινε πραγματικά αηφορία. Το ίδιο για το θέμα της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής των φορολογικών παραδείσων. Καλό είναι που σημειώνεται κάποια κίνηση, αλλά δεν αρκούν αυτά τα πράγματα, το γνωρίζουν όλοι. Οι χώρες οι οποίες εξακολουθούν να αντιδρούν, ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν. Αν όμως εξακολουθήσουν να υπάρχουν τρίτες χώρες οι οποίες δεν συνεργάζονται, επειδή και εγώ βάζω αναγκαστικά τα ρήματά μου στο τέλος της φράσης, έχω να σας πω και για την ανεργία. Δώστε μου ακόμα λίγα δευτερόλεπτα. Ελπίζω στην νομοθετική διαδικασία να μην αποδυναμωθεί η προσπάθεια για την αντιμετώπιση ανεργίας. Αυτά όμως τα μηνύματα να τα δώσετε κυρίως στους υπουργούς του Συμβουλίου, που αυτοί είναι που παίρνουν τις αποφάσεις. Και κατά τα άλλα γνωράζετε πολύ, γνωρίζετε πολύ καλό ότι τα 6 δισεκατομμύρια δεν αρκούν για τίποτα. Σύμφωνα με την Διεθνή Οργάνωση Εργασία χρειαζόμαστε τουλάχιστον 21 δισεκατομμύρια. Ο κύριο Βαντεστούπ τώρα από πλευρά μη εγγεγραμμένων για δύο λεπτά. Και με τον κύριο Βαντεστούπ ολοκληρώνεται ο γύρος των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των διαφόρων ομάδων. Έχετε δύο λεπτά κύριε Βαντεστούπ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν μιλώ εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων, είμαι μέλο των μη εγγεγραμμένων. Πρόεδρε, δεν θέλετε να σήμερα για τους μισθούς των ευρωϊπαλλήλων. Όπως είπε ο κύριος Σούλτ την περασμένη εβδομάδα, ε, μειώνεται η υποστήριξη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Στον Αδύρι είναι. Ο πρόεδρος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όμως δεν λέει τι τρέχει. Ε, εγώ θα σας πω ο κόσμος ε, έχει βαρεθεί τις Βρυξέλλες, έχει βαρεθεί το ευρώ, το 3%, τα ανοιχτά σύνορα και ε, πρώην πολίτες Ανατολικής Ευρώπης που έχουν κατακλείσει τη Δυτική Ευρώπη. Με δύο λόγια ο κόσμος έχει βαρεθεί την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ηγέτες της, ε, διότι δεν ξέρουν ιδέα, δεν έχουν τι συμβαίνει στους απλούς ανθρώπους. Πού οφείλεται αυτό? το ευρώ έχει ε, αποδυναμώσει τις χώρες ε, και τις αναγκάζει να κάνουν μεταρρυθμίσεις ε, με στρατιές ευρωϊπαλλήλων. Ο κύριος Τίμερμανς Ολλανδός Υπουργός Εξωτερικών με εντολή ε, του Ολλανδικού Κοινοβουλίου δεν πρόκειται να γυρίσει στη χώρα του εάν δεν του πούνε πόσοι είναι οι Ευρωπαίοι υπάλληλοι που κερδίζουν περισσότερα από τον Πρωθυπουργό της Ολλανδίας το χρόνο. Λοιπόν, ε, έχω ρωτήσει επανειλημμένα, γραπτός, αλλά οι ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπεκφεύγουν. Ο ε, Ολλανδός ε, Εξωτερικών δήλωσε ήδη ότι θέλει να γνωρίζει τι γίνεται. Πάνω από 3.000 ευρωϋπάλληλοι κερδίζουν μεικτά περισσότερο από τον Ολλανδό Πρωθυπουργό βάλε και τα επιδόματα και τα λοιπά έξτρα ε, ε, εισοδήματα, αυτοί υπερβαίνουν τις 10.000 παρακαλώ. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα σήμερα. Αυτή ε, την ενημέρωση ζητήσαμε και δεν την παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορείτε στο Κοινοβούλιο να ενημερώσετε, να διαβιβάσετε την πληροφόρηση αυτή, κύριε Μπαρόσο. Επαναλαμβάνω, πόσοι ευρωϊπάλληλοι που εργάζονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν πάνω από 144.000 στο χρόνο ε, με όλα τα επιδόματα τέκνων, ε, αποδημίας και πάει λέγοντας. Και ε, ο, ο φόρος ελεγγύης του 15% είναι. πάνω από 10.000 ή όχι. Η απάντηση είναι απλή. Κάπου στην Ευρώπη δεν μπορεί κάποιος να απαντήσει ένα κουμπί για να μας τα στείλει αυτά. Ο απλός πολίτης αυτέ τις απαντήσει θέλει. Παρακαλώ να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ ο Πρόεδρος. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά στον Πρόεδρο του Συμβουλίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει και ένας γύρος ομιλητών, ένας από κάθε ομάδα με την αντίστροφη σειρά από τη μικρότερη προς τη μεγαλύτερη. Ο κύριος Μπαρός έχει πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις που ε, ήταν εγγεγραμμένε στη μερίσια διάταξη, δηλαδή που αφορούσαν θέματα που συζητήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν πρόκειται να μπω σε άλλα θέματα, έστω και αν είναι πολύ ενδιαφέροντα. Με μεγάλη χαρά να απαντήσω γραπτό αν επιθυμείτε ε, και αν τις ε, θέσετε τις ερωτήσεις σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα σημερινά θέματα που μας απασχολούν. Είναι η φορολογία και η ενέργεια. Και μερικά άλλα. Παρακαλώ ε, σύντομα να απαντήσω στα σχόλιά σας. Σε ό,τι αφορά τα όσα είπαν οι κυρίες Τσίμερ και Χάρμς, δεν συμφωνώ ότι αλλάζουμε παράδειγμα. Δηλαδή, δεν συμφωνώ ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που απεμπολούμε την ε, προσήλωσή μας στη βιωσιμότητα και την αηφορία. Τι συμβαίνει έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγέ και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε στο παγκόσμιο ενεργειακό τοπίο και είμαστε υποχρεωμένοι να το λαμβάνουμε υπόψη αυτό στη χάραξη πολιτικής σήμερα. Και η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περί αυτού εστράφει. Ε, ο ενεργειακό χάρτη σήμερα δεν είναι ο ίδιο με εκείνο πριν από 5-6 χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολείποτε μάλλον όλων όσων έχει προτείνει για ως πολιτική και για την ενέργεια και για το κλίμα. Και δεν θα πρέπει να ενδώσουμε. Είχαμε ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής παγκοσμίω. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ε, καταλάβουμε ποιοι είναι οι νέοι περιορισμοί στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Η παγκόσμια εκμετάλλευση νέων πόρων, ιδιαίτερα το ε, σχισολιθικό αέριο στι Ηνωμένε Πολιτείε έχει δώσει τεράστια όθηση στι παγκόσμιε αγορέ. Και αυτό έχει αντίκτυπο και στι διαφορέ και στη δημολόγηση τη ενέργεια, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα στην Ευρώπη βλέπουμε χαμηλέ επενδύσει, ακριβώ λόγω τη οικονομική κρίση. Ε, το ατύχημα στη Φουκουσίμα επηρέασε κατά τεράστιο βαθμό τι επιλογέ ε, ω προ την ενέργεια σε ορισμένα κράτη-μέλη και βεβαίω έχει επιπτώσει και στα βήματα που παίρνουν ε, και κάνουν οι κυβερνήσεις. Και ένα τελευταίο, χωρίς να είναι αυτό λιγότερο σημαντικό, βλέπουμε στην όλη ε, εσωτερική αγορά να γίνονται ειδικέ επιλογές από τα κράτη-μέλη που είναι εμπόδιο για την ανταγωνιστικότητα. Και αυτό οδηγεί μάλλον σε κατακαιρματισμό στην Ευρώπη περισσότερο από ότι σε ολοκλήρωση. Ε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκανα την αρχική παρουσίαση για αυτή τη συζήτηση και τους είπα ότι δεν θα πρέπει να ε, παρετηθούμε. Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Ε, ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς, ευφυείς υποδομές, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και επίσης ε, προώθησα και αυτή την ιδέα. Στις Ηνωμένε Πολιτείες γίνεται επανάσταση ως προς το ε, σχιστολιθικό. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε την ενεργειακή μας επανάσταση στην Ευρώπη. Και νομίζω αυτό συνάδει πάρα πολύ με την ατζέντα και το πρόγραμμα αηφορίας. Με περισσότερες επενδύσεις και στις ανανεώσιμες βέβαια, αλλά εκεί χρειάζεται να έχουμε μία διεθνή φωνή. Ε, αυτές είναι προτάσεις που έχουμε κάνει. Ε, καλωσορίζω και χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατανόησε το ρόλο κλειδί ε, που έχει το πλαίσιο για το 2030 για το κλίμα και την ενέργεια για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε υποδομές. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2013 το Μάρτιο θα εξετάσει τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθοδήγηση και οι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάντα ευπρόσδεκτε. Το συζητούμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω παρακαλώ να το καταλάβουμε. Συζητούμε ποια ε, ε, μπορεί να είναι η πολιτική και το πλαίσιο μετά το 2020. Και όταν συζητούμε αυτά τα θέματα με τη βιομηχανία παντού στην Ευρώπη και εκείνοι ζητούν ένα πλαίσιο για να μπορούν να κανονίσουν την πορεία του, τι επενδύσει του με μια ασφάλεια Εξου, λοιπόν, ε, η αηφορία, η ανταγωνιστικότητα και η ε, ασφάλεια εφοδιασμού. Να πω δύο λόγια για το σχιστολιθικό αέριο για να απευθευθούν παρεξηγήσεις. Όπω γνωρίζετε, τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για τι βασικέ αποφάσει για το ενεργειακό του μείγμα και αυτό αφορά και τη διερεύνηση και την ε, παραγωγή, εξόριξη και του σχιστολιθικού αερίου. Αυτό παραμένει ενισχύει. Ταυτόχρονα όμω, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι τέτοιες δραστηριότητες ε, συνάδων με το ευρωπαϊκό δίκαιο και το περιβαλλοντικό και της ε, δημόσιας υγείας. Ε, εμείς θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι οι κανόνες του παιχνιδιού είναι ήδη παντού σε όλη την Ευρώπη εξασφαλίζοντας στο κοινό ότι υπάρχουν ε, τα ε, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής τους. Ε, αυτό που χρειάζεται λοιπόν είναι ένα πλαίσιο για ασφαλή εξόριξη συσσωληθικού αερίου και αυτή η πρόταση θα έρθει μέχρι το τέλος του έτους εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα με ανοιχτή διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους και τα κρατη και τη βιομηχανία και την κοινωνία των πολιτών. Αυτά θα ήθελα να σας πω για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, δεν έχουμε αλλάξει παράδειγμα, αλλά τουλάχιστον εγώ έτσι εξέλαβα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το πνεύμα, διότι συμμετείχα και στις συζητήσεις αυτές. Πλην όμως ε, είναι γεγονός ότι δόθη μεγαλύτερη έμφαση στο θέμα της ανταγωνιστικότητας. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να το εκλαμβάνουμε ως πίεση. Ή ότι είναι ε, κάτι ε, το οποίο αντιτίθεται στη δέσμευσή μας για την αηφορία και τη βιωσιμότητα. Είναι νέα τα δεδομένα όμως ε, από την οικονομική πίεση για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, γιατί αλλάζει το παγκόσμιο τοπίο, είπαμε, στην ενέργεια. Τώρα, ένα γενικότερο σχόλιο, γιατί οι περισσότερες ερωτήσεις ε, απευθύνθηκαν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με την φορολογία. Αλλά να αναφέρω αν κατάλαβα καλά ο Πάολο Χαζέλ πρότεινε μια ε, ομοιόμορφη ε, φορολογία στην Ευρώπη. Δεν είναι δυνατόν όμως αυτό και πιθανότατα δεν είναι καν επιθυμητό. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, ανταγωνιστική Ευρώπη με διαφορετικά φορολογικά συστήματα, αλλά χρειαζόμαστε και αυτό ισχύει, ιδιαίτερα όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή φορολόγηση και πρέπει να, να αποφύγουμε αυτή την πρακτική της επιθετικής φορολογικής, του επιθετικού φορολογικού ε, σχεδιασμού. Πιο πολύ συνοχή, όπως πρότεινε ο Πάολο Ραζέλ, αλλά φεύγοντας την ε, ομοιομορφία που μπορεί να φέρει άλλα προβλήματα όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά μας. Και έπειτα η, ανησυχία σε σχέση με τις πιο φτωχές περιοχές και τις πιο ευάλωτες περιοχές σήμερα λαμβάνεται υπόψη από την Κομισιόν ε, όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές μας για τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Ε, κάνουμε θετικές διακρίσεις. Υπάρχουν δυνατότητες για φορολογικά κίνητρα προς τις πιο ευάλωτες χώρες και περιφέρειες. Και εδώ σίγουρα θα το επιβεβαιώσουμε στην αναθεώρηση γιατί είναι και θέμα ισότητας και δικαιοσύνης. Επίσης θα ήθελα να τονίσω τα όσα είπε ο πρόεδρος Βαναρομπόη και εγώ, αλλά και άλλοι όσον αφορά το θέμα της ανεργίας των νέων. Και είμαστε πολύ ειλικρινείς σε αυτό το θέμα. Πρόσφατα βλέπουμε μια, ένα πολλαπλασιασμό πρωτοβουλειών για το θέμα αυτό και πραγματικά καλωσορίζω τις πρωτοβουλίες αυτές. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι οι πρωτεύουσε στην Ευρώπη που παλιότερα δεν ήταν τόσο προσιλωμένες σε αυτό το θέμα, τώρα ε, εργάζονται δραστήρια και δίνουν όχι μόνο πολιτική δέσμευση αλλά και εμπειρογνωμοσύνη, διότι για να σας δώσω ένα παραδείγμα στη Γερμανία υπάρχει πολύ μεγάλη εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις δραστήριες εργατικές πολιτικές, κυρίως μετά από την ενοποίηση της Γερμανίας. Και μπορώ μόνο να καλωσορίσω και να συγχαρώ αυτές τις πρωτεύουσε που τώρα εργάζονται ενεργά δραστήρια ώστε να δώσουν περισσότερα και σε σχέση με τη διακυβερνητική συνεργασία ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που το χρειάζονται περισσότερο. Τώρα όμως αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται εις βάρος των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων και των προσεγγίσεων της ευρωπαϊκής κοινότητας. Και αυτό είναι το θέμα. Και να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Το 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 11 με συγχωρείτε, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με εγγυήσει ε, που στόχο είχαν ένα συμπληρωματικό δημοσιονομικό μέσο για να διαχειριστούμε το κοινωνικό ταμείο. Αυτή η πρόταση απορρίφθηκε και τον Νοάριο ε, λόγω τη Γερμανία, Δανία, Σουηδία και του Ηνωμένου Βασιλείου για τις θέσεις του. Το απέρριψαν. Τώρα όμω η ιδέα που έρχεται ε, είναι ε, αυτό το New Deal ε, είναι πολύ κοντινό να φέρουμε δηλαδή την ιδέα εγγυήσεων μέσω ευρωπαϊκών μέσων. Ωραία, αλλά δεν θα ήταν καλύτερα να το είχαμε από νωρίτερα, να είχαμε αυτές τις εγγυήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και αυτό είναι το σημείο στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε. Επειδή θέλω να είμαι πολύ ειλικρινή μαζί σα, ο πολλαπλασιασμό νέων πρωτοβουλειών, όταν δεν υπάρχει ακόμα εφαρμογή των παλιών πρωτοβουλειών, δεν είναι αξιόπιστη. Και γι' αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει για την εφαρμογή των αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί, όπω η εγγύηση τη της που διοθετήθηκε ε, πολύ σύντομα από τα κράτη-μέλη. Μάλιστα η πρόταση της Κομισιόν με πολύ στεναρή στήριξη από το Ευρωκοινοβούλιο. Ας εφαρμόσουμε αυτό που ήδη έχουμε υιοθετήσει. Ας είμαστε σοβαροί. Ας, ας δώσουμε αποτελέσματα. Και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ συμφωνώ με τις επικρίσεις αυτές που ακούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πολύ συχνά λαμβάνουμε αποφάσεις αλλά μετά κολλάμε στην εφαρμογή. Και οι πολίτες δεν βλέπουν τη μετάφραση των αποφάσεων αυτών στην πράξη. Πολλές φορές μάλιστα λαμβάνονται σε πολύ ψηλό επίπεδο, σε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν τις βλέπουν όμως αποφάσεις αυτές να επηρεάζουν την καθημερινά του ζωή. Θα πρέπει να σας πω ότι το πνεύμα όμως υπάρχει πια και ότι πρέπει να φτιαχτεί αυτή η συνένεση για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου που πιστεύω θα λάβει πολύ σημαντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει τώρα ο κ. Βαρόν Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για να απαντήσει στις ερωτήσεις και τα σχόλια των συναδέλφων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Γράψαμε στην ημερήσια διάταξη σήμερα δύο θέματα. Την ενέργεια και τους φόρους. Αυτά είναι θέματα που παραμένει πάρα πολύ σημαντική η εθνική αρμοδιότητα για την ενέργεια, το λεγόμενο ενεργειακό μείγμα βοηθάει την εθνική ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό. Ή παραμένει ε, εθνική αρμοδιότητα. Ε, η φορολογία είναι θέμα ε, που παραμένει στην ομοφωνία. Δηλαδή, όταν συζητούμε για αυτά τα θέματα βρισκόμαστε σε λίγο μειονεκτική θέση γιατί η κύρια αρμοδιότητα και εξουσία παραμένει σε εθνικό επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν μπορούμε ουσιαστικά να λύσουμε το πρόβλημα της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής. Ε, δεν μπορούμε να λύσουμε τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς τη τιμολόγηση της ενέργειας, τον εφοδιασμό ε, μόνο αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν πλήρη επίγνωση της σημασίας του ευρωπαϊκού επίπεδου και σε αυτά τα θέματα, γνωρίζοντας ταυτόχρονα τους περιορισμούς που έχουμε λόγω κατανομής των αρμοδιοτήτων. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Ε, πρώτο σχόλιο αυτό. Δεύτερον, παρά το γεγονός ότι πολλοί ε, επιμείνατε να υπάρξει μεγαλύτερη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να καταλάβουμε, το ξέρω το γνωρίζετε, θα ήθελα απλώς να το υπενθυμίσω, ότι ακόμα και πριν την ε, χρηματοπιστωτική κρίση υπήρχαν πολλές διαφορές και αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Μιλώ για τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Ε, κοιτώ τα αριθμητικά στοιχεία για την παραοικονομία για τη μαύρη εργασία είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα η εικόνα. Άρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο βεβαίως θα πρέπει να δράσουμε, αλλά αυτό δεν αποκλείει τις δράσεις που μπορούν να αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο με τρόπο πάρα πολύ πιο επεμβατικό, με θεαματικά αποτελέσματα σε ορισμένες χώρες. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε επίγνωση της σημασίας του ευρωπαϊκού επίπεδου, θα πρέπει ακόμα περισσότερο να γνωρίζουμε ε, πόσο σημαντική είναι η δράση σε εθνικό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενέργεια των νέων. Πολύ πριν τη χρηματοοικονομική κρίση υπήρχαν μεγάλες διαφορές επίσης ως προς την ανεργία των νέων. Και εκεί η δράση σε επίπεδο κράτους μέλους μπορεί να ε, αποδειχθεί αποτελεσματική. Εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο σε επίπεδο κρατών μελών. Δεν θέλω και πάλι να δώσω την εντύπωση ότι ε, δεν ε, υπάρχει καμία δυνατότητα δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει. Αλλά θα ήθελα να εμείνω στο γεγονός ότι απαιτούνται δράσεις σε διάφορα επίπεδα. Τρίτο σχόλιο. Χαίρομαι που μιλήσαμε για τη φοροδιαφυγή και για τη φοροαποφυγή. Ορισμένοι από εσάς αναφέρουν το θέμα αυτό χρόνια ολόκληρα. Αλλά διαπιστώνω ότι από τότε που εγγράφηκε στην διάταξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτό το θέμα, έχει επιταχυνθεί η συζήτηση. Και έχει ενταθεί επίσης. Ε, αυτός ήταν ο στόχος άλλωστε. να συζητηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αυτό ε, ενθάρρυνε και τους Υπουργούς Οικονομικών να λάβουν πρωτοβουλίες, αλλά και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να λάβουν αποφάσεις. Και αποφάσεις ελήφθησαν. Ποιος θα έλεγε, έστω και πριν από λίγους μήνες, ότι ήδη τον Ιούνιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα καταθέσει οδηγία για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εισοδημάτων. Καλά, βεβαίως, ήδη ε, υπήρχαν στο παρελθόν πρωτοβουλίες για τα εισοδήματα από καταθέσεις και από ταμείευση, αλλά για όλα τα εισοδήματα, για μια ευρεία έτσι, ε, γάμα εισοδημάτων, είναι πρώτη φορά. Ε, βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια καμπή πλέον. Και βεβαίω αυτό βοηθήθηκε και από την πρωτοβουλία των πέντε Υπουργών Οικονομικών. Αλλά δεν θέλουμε αυτό να παραμείνει σε επίπεδο πρωτοβουλίας ε, ορισμένων χωρών που θα οδηγηθεί σε εμπλοκή, αλλά να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο 27 κρατών, προσεχώς 28. Ε, θα προχωρήσουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη τον Ιούνιο ε, τα θέτει πρόταση. Επιτέλους, επίσης έχουμε εντολή για διαπραγμάτευση με την Ελβετία και τις υπόλοιπες χώρες. Μετά από χρόνια και χρόνια συζητήσεων, επιτέλους έχουμε εντολή. Ταυτόχρονα όμως είπαμε, στο σημείο Β, του 10 των συμπερασμάτων και παραθέτων, λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρων και ε, υπόψη επίσης και της αναθεωρημένης οδηγίας για τα εισοδήματα από καταθέσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε να εγκριθεί πριν το τέλος του έτους η πρόταση αυτή. Τέλος παράθεση. Βεβαίως υπάρχει εκεί μια σχέση, αλλά μπορεί να προχωρήσει το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά την οδηγία για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από καταθέσεις, έτσι ώστε πριν τα τέλη του έτους να υπάρχει συμπέρασμα, να έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η παράγραφος Β συζητήθηκε πολύ και με τρόπο πάρα πολύ συγκεκριμένο και πραγματικά εννοεί αυτό που λέει. Δηλαδή, είναι πολύ ευρύτερη από ό,τι ορισμένοι θεωρούν ή υποπτεύονται. Έγινε λοιπόν αυτή η ακαμπή. Ορισμένοι από εσά μίλησαν για μια πρόταση που έχει στόχο να τροποποιήσει τις οδηγίες για την ε, ε, δημοσίευση μη οικονομικών πληροφοριών ε, σε σχέση με τη διαφοροποίηση στην οποία προβαίνουν ορισμένε μεγάλες εταιρείες και μεγάλοι όμιλοι αναχώρα. Για τις τράπεζες, και αυτό είναι ευρέως γνωστό, έχουμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο χάρη στην ε, οδηγία ε, για τις κεφαλαιακές απαιτήσει 4. Ε, ήδη έχουμε φτάσει στη διαφάνεια. Μιλούμε για μια οδηγία που περνά από, τη διαφοροποίηση και τα μη χρηματοοικονομικά, αλλά στο μεταξύ έχει γίνει μια συμφωνία στο τριμερή διάλογο ως προς την διαφάνεια και τη λογοδοσία. Και μάλιστα αυτή αναφέρεται και στα συμπεράσματα. Εάν οι συνομοθέτες ε, συμφωνήσουν για τροπολογίες που ε, θα αυξήσουν έτσι περαιτέρω τη διαφάνεια, κανείς δεν τους εμποδίζει να το υιοθετήσουν και να ε, βρουν και μια μορφή συμβιβασμού με το Συμβούλιο. Ε, σχέση με τους φορολογικούς παραδείσους θα ήθελα να αναφέρω μόνο που δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή. Ε, σας παραπέμπω στις δηλώσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού πριν από λίγες εβδομάδες που ανακοίνωσε μεγαλύτερη διαφάνεια των καταθέσεων και των λογαριασμών σε ε, εδάφη ε, όπως ονομάζονται ε, είναι εξαρτημένα από το βρετανικό στέμα και υπεράκτιες βρετανικές κτίσεις. Παντού λοιπόν σε όλα αυτά τα θέματα καταφέραμε όχι απλώς να κάνουμε πρόοδους αλλά και ουσιαστικές πρόοδους, καμπή κάθε φορά αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ε, για ένα όσο γίνεται ευρύτερο φάσμα εισοδημάτων. Αυτό είναι πραγματική επανάσταση ε, στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των φορολογικών απατών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως όλα αυτά θα πρέπει να υλοποιηθούν. Αλλά δεν μπορεί κανείς ταυτόχρονα και να αποφασίζει και να εκτελεί. Ε, δεν θα πρέπει να μας... Αλλά ελπίζω ότι θα μας ελέγξετε και όλα ως προς αυτό, ε, με, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ε, σας ε, αναφέρουμε τα σημεία που έχουμε επιτύχει πρόοδο. Στο σημείο 11 αναφέρεται αυτό ρητά. Μέχρι το Δεκέμβριο 2013 σε τακτά επαναλαμβάνω χρονικά διαστήματα θα αξιολογούμε πού βρισκόμαστε στην εκτέλεση των ιδίων μας των συμπερασμάτων. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε ευρύτατα για την ενέργεια, δεν θα αναφερθώ εγώ ούτε θα επιμείνω σε αυτό. Να πω μόνο το εξής. Όταν ορισμένοι λέγουν ότι η διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη είναι λίγα χρήματα, μόνο 5 δις, θα μπορούσαν να είναι περισσότερα, πάντα θα μπορούσαν να είναι περισσότερα. Τα 6 δις που προβλέψαμε για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας και αυτή είναι ε, μικρή ε, προσπάθεια, είναι μικρά τα ποσά. Αλλά εγκρίνουμε πρώτα τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Κάποιο φωνάζει από κάτω, εξαρτάται από το Συμβούλιο. Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά θα πρέπει να ε, συμφωνήσουμε για ένα πολιετές πλαίσιο δημοσιονομικό. Αν μη τι άλλο, τότε θα έχουμε αυτά τα 5 δισεκατομμύρια για τη διευκόλυνση συνδέοντας στην Ευρώπη. Και αν μη τι άλλο, θα έχουμε τα 6 δις για την ανεργία των νέων. Αλλιώς δεν θα έχουμε ούτε αυτά. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε για να ε, υπάρξει κοινοτικό προπολογισμό για την περίοδο 2014-2020. Για την ανεργία των νέων, όπω και ο πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χαίρομαι για τι νέε πρωτοβουλίε. Ήδη έχουμε εργαστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δεν αρκεί όμως αυτή η προσπάθεια, διότι υπάρχει τώρα και μια νέα αποστολή που είναι αδιαμφισβήτητη η επιτυχία μας, η εξασφάλιση της σταθερότητας της Ευρωζώνης. Κανείς δεν αναφέρεται πλέον στην κατάρρευση της Ευρωζώνης ή την, το θάνατο του ευρώ. Ε, τώρα όμως θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να καταπολεμηθεί η οικονομική κρίση και η ενεργεία και οπωσδήποτε η ενεργεία των νέων. Λοιπόν, τον Ιούνιο ε, θα γίνει μια ενημέρωση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τι μπορούμε να κάνουμε σε εθνικό επίπεδο. Πολλές είναι οι κυβερνήσει και τα κοινοβούλια που ήδη εξήγηλαν πρωτοβουλίε, αλλά τι μπορούν να πράξουν και οι κοινωνικοί εταίροι, διότι και εκείνοι φέρουν ευθύνη. Είμαστε υπερήφανοι ε, για το σύστημα κοινωνικής διαβούλευσης που έχουμε στην Ευρώπη, αλλά και σε περίοδο κρίσης και το σύστημα των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να είναι παραγωγικό και περιμένω μια συνεισφορά από πλευρά του στις επαφές που έχουμε. Έτσι λοιπόν να υπάρχει μια γενική κινητοποίηση ε, σε όλα τα επίπεδα κατά της ανεργίας των νέων. Και ελπίζω να επανέλθουμε τον Ιούνιο για να σας αναφέρουμε τα πεπραγμένα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και να μην επιδεικνύουμε μόνο πολιτική βούληση αλλά και πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακολουθούν τώρα οι υπόλοιποι ομιλητές, ο τελευταίος γύρος, με την αντίστροφη σειρά όπως σας είπα, από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη ομάδα. Θα έχετε πολύ λίγο χρόνο όλοι σας. Ένα λεπτό παρακαλώ να τον τηρείτε. Αλλιώς οι τελευταίοι δεν θα προλάβουν. Και θα μείνουμε οι τρεις μας, αν παραμείνουν οι δύο πρόεδροι. Δεν θα έχει μεγάλη προσέλευση η ε, συνεδρίαση. Ο κύριος Βαντερστούπ. Δεν με εκπλήσει που αρνείται ο κύριος Μπαρόζο να απαντήσει αυτά που ρώτησα για τους ευρωμισθούς. Αυτό είναι το στάνταρ αντανακλαστικό όταν δεν του αρέσουν οι ερωτήσεις. Είναι ανόητα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει το θέμα ε, της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Εκεί εμπίπτουν οι φοροδιαφυγές των ευρωϊπαλλήλων στην ε, σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην ιστοσελίδα. Γιατί δεν υποστηρίζετε αυτά, γιατί δεν μας λέτε πόσοι είναι οι υπάλληλοι που κερδίζουν περισσότερα από τον ίδιο μας τον Πρωθυπουργό. Λέτε να σας κάνω γραπτή ερώτηση, τρεις φορές το έχω ρωτήσει. Ε, και ε, δεν θα απαντήσετε, δεν έχετε δεΐς, διότι φοβάστε τους πολίτες γιατί με αριθμητικά στοιχεία μπορούμε εμείς να σας καταγγείλουμε, φοβάστε μήπως θυγούν τα φιλαράκια σας, φοβάστε τη διαφάνεια, φοβάστε τη γνήσια δημοκρατία και όχι την εικονική ψευδοδημοκρατία που συνιστά σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, Πρόεδρε, και τελείωσα. Η κυρία Τσίμερ, για ένα λεπτό. Ακόμα και εάν έχουμε διαφορές αντιλήψεων, ας προσέχουμε λίγο το τόνο της φωνής μας και το ύφος. Δεν συμφωνώ μαζί σας σχετικά με, το, με την αλλαγή παραδείγματος. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει κανείς να διαβάζει και ανάμεσα στις γραμμές και βεβαίως να μιλεί και για όλο το σύνολο των θεμάτων. Όταν μιλείτε για μείωση του κόστους, δεν εννοείται μείωση του κόστους υπέρ της κοινωνίας για να μπορέσει να αλλάξει και η πορεία αυτής της κρίσης χρέους, αλλά μιλείτε πάντα μόνο για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Επομένως, οι στόχοι και οι ομάδες ανθρώπων δεν φτάνεται σε αυτούς με αυτή την εξοικονόμηση που προτείνεται. Και μόνο μια σύντομη φράση για την ανεργία των νέων. Ακόμα και αν οι χώρες μέλη οφείλουν να ξεκινήσουν δικές τους πρωτοβουλίες, θεωρώ ωστόσο ότι είναι σημαντικό το Συμβούλιο και τα όργανα της Ένωσης να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους, δηλαδή εγγύηση υπέρ της νεότητας, δηλαδή τα χρήματα, τουλάχιστον αυτά τα οποία έχετε υποσχεθεί, πραγματικά να τεθούν στη διάθεση του ε, στόχου αυτού και να μην χαθούν μέσα σε ένα παζάρι χωρίς να γίνει τελικά τίποτα το Ευχαριστώ για ένα λεπτό. Ο κύριος Βλόσοβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι ηγέτες της Ένωσης Έφεραν το θέμα της ενέργειας, είναι ένα μεγάλο ζήτημα και ένας τρόπος για να υποστηριχτεί η ανάπτυξη και η απασχόληση. Είναι πολύ σημαντικό η ενέργεια να καταστεί πιο προσιτή, φθηνότερη από ό,τι τώρα, γιατί κοστίζει το διπλάσιο από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Δυστυχώς η οικονομία της Ευρώπης υποφέρει από την πολιτική μας για το, από το, για το τις εκπομπές διοξίδιου του άνθρακα και αυτό εμποδίζει και τη διαδικασία βιομηχανοποίησης της υπήρου μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυηθεί την ε, πάρκια ανεφοδιασμού σε ενέργεια για τα νοικοκυριά και τις ε, επιχειρήσεις ε, και επίσης ανεφοδιασμό σε προσιτή ενέργεια. Και αν τα συμπεράσματα αυτά τεθούν σε εφαρμογή, εξακολουθεί να υπάρχει επικράτηση της κλιματικής πολιτικής επί της ενεργειακής. Μάλιστα τελικά θα καταφέρουμε το αντίθετο από αυτό που επιθυμούμε. Η ενέργεια θα καταστεί ακόμα πιο ακριβή, η βιομηχανία μας λιγότερο ανταγωνιστική και θα αυξηθεί και το κόστος για τα νοικοκυριά. Θα ήταν κρίμα να στείλουμε την, την ήπειρό μας στο βάραθρο. Ευχαριστώ. Το προνόμιο που έχει αυτή η αίθουσα σε σχέση με την Ολομέλεια είναι ότι δεν έχουν κουμπί SOS να πατήσουν οι διερμηνείς όταν τρέχετε τόσο πολύ. Και δεν με αγχώνουν με το δικό τους άγχος. Ε, για ένα λεπτό τώρα, κύριε Σκάλανε. Thank Κύριε Πρόεδρε, Καταρχήν για την ενέργεια, ε, ελπίζω πως και η κυρία Τσίμερ εδώ θα δεχτεί πως όντω υπήρξε μια αλλαγή πορείας στην πολιτική ενέργεια μας, γιατί κατά τη γνώμη μου θα ήταν αδύνατο να έχουμε συγκεκριμένη οικονομική ανάκαμψη με τα κόστη ενέργειας διπλάσια από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος ε, του ανεπτυγμένου κόσμου, για να μην ε, πάμε πίσω στις σπηλιές. Και Α, τώρα, όσον αφορά τη φορολογία, αν θέλετε να παρακμάσει η ευρωπαϊκή οικονομία, ναι, ε, ε, να αρμονίσετε τη φορολογία μας. αν θέλετε να μπούμε και πάλι στην πορεία του ανταγωνισμού, ο, ο μόνος στεναρός ε, του φορολογικός ανταγωνισμός θα βοηθήσει. Κοιτάξτε στον κόσμο τι συμβαίνει, κοιτάξτε που υπάρχει επιτυχία. Είναι τα μέρη όπου υπάρχουν τα χαμηλότερα ποσοστά άμεσης φορολογίας. Ε, δείτε, το, δείτε το πρακτικά το θέμα, δείτε πώ θα έρθει η ανάκαμψη, η έξοδο από την ύφεση και όχι πώ θα ομοσπονδοποιήσουμε τι φιλοδοξίες φιλοδοξίες μα και να χρησιμοποιήσουμε ε, αυτού του τρόπου για να προωθήσουμε τις ατζέντε ορισμένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κάλαναν και τώρα για ένα λεπτό επίση η κυρία Ρεμπέκα Χάρμ. Äh, ε, γύρομαι τώρα πλέον ως ε, εκπρόσωπος της ομάδας των ανθρώπων των σπηλαίων, διότι έτσι μας αποκάλεσε προηγουμένως ο κ. Κάλαναν. Εγώ θα ήθελα να έχω μια επισκόπηση των τιμών της βιομηχανικής ενέργειας σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, ποια είναι η επιχείρηση εκείνη η οποία κατέρευσε λόγω των τιμών ενέργειας που ζητούμε εμείς. Έχουμε τόσες πολλές εξαιρέσεις υπέρ της βιομηχανίας. Έχουμε διανύμει όλα τα πιστοποιητικά δωρεάν. Έχουν πνιγεί στα πιστοποιητικά, ενώ για τα αέρια θερμοκηπίου. Και όμως δεν έχει λειτουργήσει τίποτα. Πού βρίσκεται λοιπόν αυτή η μεγάλη τραγωδία της ε, βιομηχανίας που είναι εντατική σε χρήση ενέργειας. Πρόκειται για ανθασμένη υπόθεση και ξεκινώντας από αυτή την εσφαλμένη υπόθεση προχωρούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό, την, υπό τις κατευθύνσεις που δίνει ο Επίτροπος Έτινγκερ σε μια υπονόμευση της πολιτικής για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Παρακαλώ και πάλι, δώστε μου διαφάνεια για τις τιμές ενέργειας, ενέργειας τις οποίες χαίρει η βιομηχανία. Ευχαριστώ, κυρία Σάρον Μπόουλς. Ε, ε, Ευχαριστώ. Πρόεδρε Βαρόμπε, είπατε ότι το Κοινοβούλιο επέστησε την προσοχή ε, στη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή από την έκθεση μου από το 2008 και του Μπενουά το 2009 για τις καταθέσεις παρόλες ε, τις φιλόδοξες ε, δηλώσεις του G20 μετά τη Σύνοδο Κορυφής του 2009 ο σχεδόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε οθούν. Μέσω του ΦΑΤΚΑ τα κράτη-μέλη τώρα δίνουν πληροφόρηση στις Ηνωμένε Πολιτείε που δεν δίνουμε στους εαυτούς μας. Ε, μετά την αντίστοιχη νομοθεσία συμφωνήσαμε χώρα προς χώρα να ε, αναφέρουμε για τις εξορρυκτικές και υλοτομικές ε, βιομηχανίες. Τα ξέρω γιατί έχω ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά δεν γνωρίζουμε καθόλου τι συμβαίνει στην Ευρώπη ε, με τον τρόπο που δίνονται τα κέρδη και που φορολογούνται. Λοιπόν, μία αναφορά αναχώρα είναι πρόσδεκτη, αλλά είναι κρίμα ε, που τώρα η οδηγία για την ε, λογοδεσία και τη διαφάνεια έχουν συμφωνηθεί ακόμα και αν δεν έχουν ακόμα ε, ψηφιστεί γιατί είναι μαζική η αντίσταση εκεί του Συμβουλίου. Ένα τρισεκατομμύριο διακυβεύεται εκεί ευρώ και οι μεγάλες επιχειρήσεις ε, πληρώνουν πολύ λίγο φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορα τεχνάσματα παρά τα τεράστια κέρδη τους. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα να δούμε τι τρέχει. Εάν οι μεγάλες εταιρείες δεν πληρώνουν φόρους, ε, δεν είναι θεμητός ο ανταγωνισμός με μικρές ντόπιε εταιρείε που φορολογούνται. Έχει γίνει καμιά ανάλυση για το πόσο βλάπτει αυτό την ανάπτυξη των μικρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Υπάρχει το επιχείρημα ότι δημιουργούν θέσεις εργασίας και φόρο εισοδήματος, ε, αλλά αυτό δεν στέκει. Ε, είναι πραγματικά απάτη. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια εκμετάλλευση. Θα πρέπει κάθε χώρα και κάθε φορολογούμενος ε, να επωφεληθεί, διότι έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Ο κύριος Μπανιέ είπε ότι θέλει κάτι ουσιαστικό γρήγορα. Ε, θα μας διαβεβαιώσετε ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε παρελκυστικές ε, τακτικές ε, στο Συμβούλιο ή θα ζητήσουν ανταλλάγματα από το Κοινοβούλιο, διότι εδώ δεν είναι θέμα στην ομοφωνία, είναι συνομοθέτη στο Κοινοβούλιο. Κρίμα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα την οδηγία για τη λογοδοσία και τη διαφάνεια. Θα πρέπει να βάλουμε ένα κεφάλαιο στην οδηγία που δεν είναι οικονομική για την οικονομική αναφορά και λογοδοσία αναχώρα. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει και στην οδηγία αυτή και να ε, είναι νομικά δεσμευτικό, να επιβάλλεται και μάλιστα εντός παρούσης θητείας. Αλλιώς είναι φρούδα ελπίδα και φρούδα υπόσχεση. Ευχαριστώ. Κυρία Μπόουλς και τώρα για τρία λεπτά και μισό η κυρία Κλέβα Κέκους. Ευχαριστώ πολύ για την πλειοψηφία των Ευρωπαίων η πληρωμή των φόρων είναι απλή υπόθεση. Κάθε χρόνο υπογράφουν την φορολογική τους δήλωση ή παρακρατεί το μισθός, ε, ε μάλλον ε, το εισόδη, ο φόρος στην πηγή του εισοδήματος. Όμως, για δύο κατηγορίες Δηλαδή οι πλουσιότεροι πολίτε και οι πολυεθνικέ χαίρουν άλλη μεταχείρισης. Η Ευρώπη χάνει χρήματα και επιτρέπει κατάχρηση των νόμων της. Και αυτές οι τακτικές διαφυγής οδηγούν σε απώλεια 1 δισεκατομμυρίου ευρώ τον χρόνο. Περισσότερο από ό,τι χρησιμοποιούμε και για το δημοσιονομικό πλαίσιο και για την υγεία σε όλη την Ευρώπη. Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήθηκε η έκθεσή μου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς καταλήξαμε στις τρεις προτάσεις. Σας παρακαλώ, σας οικετεύω κύριε Μπαρόσο. Διαβάστε τις προτάσεις αυτές. Προτείνουμε ξεκάθαρα μέτρα για το πώς θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Δεν χρειαζόμαστε νομικά μη δεσμευτικές συστάσεις. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη στρατηγική φορολογική εναρμόνιση με ένα συγκεκριμένο σημαντικό στόχο που δεν αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Πρέπει το κείμενο να είναι δεσμευτικό μέχρι το 2020 και να έχει εγκριθεί και να έχει τεθεί σε ισχύ. Τι μπορούμε να αναμένουμε λοιπόν κύριε Μπαρόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις επόμενες εβδομάδες, μήνες και μέχρι τέλους του έτους το Συμβούλιο είναι λιγότερο φιλόδοξο από την Κομισιόν. Και τα δύο αυτά όργανα είναι λιγότερο φιλόδοξα από το Κοινοβούλιο. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε τα όσα λέτε. Μπορούμε να περιμένουμε μια πρόοδο από τις συστάσεις που έγιναν πέρσι. Στα τέλη του περσινού έτους η στάση της Κομισιόν ήταν πολύ ρεαλιστική. Βέβαια, η Κομισιόν δεν προχώρησε αρκετά. Το Κοινοβούλιο προχώρησε. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω εάν η Κομισιόν προτίθεται να μελετήσει σε βάθος τις προτάσεις μας και αν μπορούμε να αναμένουμε κάπως περισσότερα από εσά. Και όχι μοναχά ένα καθαρά τεχνικό σχέδιο δράσης. Μετά από τόσα χρόνια όπου δεν συζητήθηκε καν η φορολογική πολιτική, είναι καλό που τώρα αρχίζουμε και τη συζητούμε. Όμως, στα συμπεράσματα που δημοσιεύσατε δεν λέτε τίποτα για την αναχέτηση της, φορο... της ε, ε, νομοθεσίας κατά της φορολογικής απάτης που δεν προχωρεί. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα από πέρσι είναι η απάτη σχετικά με τον φόρο προσθέμενης αξίας. Αυτό είναι από τα πιο σημαντικά. Θα ήθελα λοιπόν να δω εάν θα προωθήσετε τις ιδέες αυτές. Και επίσης η οδηγία για την φορολόγηση των καταθέσεων ελπίζω να υπάρξει μέχρι τέλους του έτους. Κύριε Βαν Ρομπόι, γιατί δεν θελήσατε να κάνετε ένα βήμα παραπέρα σε αυτόν τον αγώνα κατά των φορολογικών παραδείσων εμείς φτιάξαμε και ορισμό, ταχθήκαμε και υπέρ Ενό μαύρου κατάλογου των φορολογικών παραδείσων, αλλά στα συμπεράσματά σα, δεν διαλαμβάνετε τίποτα σχετικό. Σας ευχαριστώ και τώρα τελευταία για τέσσερα λεπτά η κυρία Σαρτόρη παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εμείς δεχόμαστε με ευνοϊκά τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ενέργεια, γιατί παρέχουν ε, έγκυρες πολιτικές προτάσεις. Θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στον ορισμό των ε, θεματικών μας στόχων, αλλά επίσης θα πρέπει να ε, αξιολογήσουμε την ανταγωνιστικότητα των τιμών που θα είναι προσιτή για τους με μονομένους χρήστες, τους ιδιώτες αλλά και για τις επιχειρήσεις. Η τιμή της ενέργειας ε, θα παραμείνει ψηλά και στο εγγύς μέλλον και δύσκολα θα μπορέσει να μας οδηγήσει στο να έχουμε τα κόστη ε, του ΙΠΑ ή άλλων χωρών. Αυτό το οποίο οφείλουμε και μπορούμε να κάνουμε είναι να περιορίσουμε όσο γίνεται περισσότερο αυτή τη διαφορά που μπορεί να, να είναι κρίσιμη για την βιομηχανική μας ανταγωνιστικότητα. Διαφορετικά θα κινδυνεύσουμε να χάσουμε την ανταγωνιστικότητα των μεγάλων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη στήριξη των πολιτών μας. Πρέπει να υλοποιηθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας, ε, ευνοώντα τις επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές που θεωρούνται απαραίτητε για το μέλλον της Ένωσης, τόσο όσον αφορά τα, ε, τα δίκτυα υποδομών για την παροχή προς την Ευρώπη, αλλά και όσον αφορά την εσωτερική, τις εσωτερικές υποδομές και τη δικτύωση. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, ωστόσο, δεν μα ικανοποιούν σε σχέση με του πόρους που τίθενται στη διάθεσή μα για όλα αυτά, αλλά ελπίζουμε πω τουλάχιστον ε, θα κινητοποιήσουν αυτές τις ε, οικονομικές δυνατότητε, όπως υποχρέωση τη σχέση, τη στήριξη τη ε, ΤΕΠ και άλλων που θα μπορέσουν να μα οδηγήσουν στο να υλοποιήσουμε αυτές τις επενδύσεις στι υποδομές. Η Ευρώπη από μόνη δεν μπορεί να αλλάξει την παγκόσμια κλιματική κατάσταση. Το 2012 ήμασταν υπεύθυνη περίπου για το 11% των παγκοσμίων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, ενώ οι εκπομπές τη Ένωση μειώνονται, αυξάνονται οι εκπομπές άλλων χωρών του κόσμου που ελέγχουν λιγότερο από ό,τι εμάς αυτή τη ε, διαδικασία. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την ε, ηγετική μας θέση όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική, αλλά γνωρίζουμε επίσης πώς οφείλουμε να διατηρήσουμε τη, σε, εν ζωή τις βιομηχανίες μας και τις θέσεις απασχόλησης για τους εργαζομένους μας. Στο πλαίσιο αυτό δεχόμαστε ευνοϊκά το γεγονός ότι συζητήθηκε έστω και σύντομα ε, μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής ενέργειας και του κλίματος σε σχέση με τον ορίζοντα 2030 το θέμα και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε για περιοχές συγκεκριμένες προτάσεις σε θέματα ενέργειας και κλίματος πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου την Άνοιξη. Θα θέλαμε ωστόσο να υπογραμμίσουμε πως η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί μετά από τους στόχους ε, τους διαπραγματευτικούς για την COP21 το 2015. Οι πολιτικές θα πρέπει να οδηγήσουν στο να μειωθεί η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και ταυτόχρονα να διώσουν τη δυνατότητα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες ενεργειακές πολιτικές, βιώσιμες και αποτελεσματικές. Αυτές οι πολιτικές θα πρέπει εξάλλου να ευνοήσουν τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, να μας καταστήσουν λιγότερο εξαρτημένους από τις εισαγωγές ενέργειας και να συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Χρειαζόμαστε να αναχαιτήσουμε τις αδυναμίες των, των πολιτικών, να αναπτύξουμε έναν ευρωπαϊκό οικονομικό μηχανισμό πιο ολοκληρωμένο που θα στηρίξει τις ανανεώσιμες ε, τεχνολογίες και θα μας καταστήσει πιο ανταγωνιστικούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε ευτυχείς για τις δηλώσεις τέλος του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, για τις ε, χώρες πηγές και για το θέμα του ενεργειακού μείγματος που παραμένει στην ε, αρμοδιότητα των κατόνοχων μελών. Θα θέλαμε όμως να θυμίσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως τα κάτι μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν είτε να περιοριστούν στη χρήση συγκεκριμένων μορφών ενέργειας τη στιγμή που η εκμετάλλευσή τους και η μεταποίησή τους επιτρέπουν ε, μια, μια αποδεκτή, έναν αποδεκτό αντίκτυπο στο κλίμα. Για την πορεία προς το 2050 επαναλαμβάνεται πως θα είναι απαραίτητε σε όλες τις τεχνολογίες με μικρή περιεκτικότητα σε άνθρακα με στόχο να, απα, να απαλλαγεί από τον άνθρακα το σύστημα της ενέργειας. Και ιδιαίτερα για την ηλεκτρική ενέργεια σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ε, που παραμείνατε και τους δύο προέδρους, Βαν και Μπαρόσο. Ολοκληρώνεται εδώ αυτή η συνεδρίαση. Πάντα ε, με ειλικρίνεια και εγκαρδιότητα ε, απευθύνεστε σε μας και θα ήθελα να σας πω μια παροιμία που λένε στη Μάντσα από όπου κατάγομαι ότι η ταπεινότητα είναι αρετή, αλλά ε, η αυταρέσκεια ε, είναι μέγα ελάττωμα ε, και αυτό δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα τέτοιους χαλεπούς καιρούς. Λοιπόν, ας πιέσουμε προς ένα δρόμο που αν πιέσουμε και μαζί προς την ίδια κατεύθυνση έχουμε μεγάλες πιθανότητες να ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια. συνεδρία συνεδρίαση.